Good morning, ladies and gentlemen. Please. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Leider ist unsere Präsidentin Frau Verheyen Δυστυχώς η πρόεδρος ε, είναι ακόμα ε, στην κίνηση και δεν έχει καταφτάσει και έτσι θα χρειαστεί να προεδρεύσω εγώ ως αντιπρόεδρος. Ε. Να ξεκινήσω λοιπόν τη συνεδρίαση και ενδεχομένως να καταφτάσει και ο πρόεδρος. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από πλευρά σας, να εγκρίνουμε το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Τα πρακτικά της 24ης Σεπτεμβρίου και της 1ης Οκτωβρίου θα τα βρείτε στα έγγραφα της συνεδρίασης. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις να κάνετε για τα πρακτικά αυτά. Δεν βλέπω να ζητάει κανεί το λόγο. Γι' αυτό θα προτείνω να θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά εφόσον φυσικά δεν εκφραστούν αντιρρήσει ε, στη διάρκεια της συνεδρίασής μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε διερμηνία στα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσαχικά, ουγγρικά, λιθανικά, λετωνικά, πολωνικά, σλοβακικά, σλοβενικά, βουλγάρικα, ρουμάνικα και κροατικά. κροατικά. Ε, ελληνικά και να μιλήσετε και να ακούσετε μπορείτε. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι η συνεδρία μεταδίδεται στο διαδίκτυο και επίσης να σας ανακοινώσω ότι αν αποφάσεις των συντονιστών της 1ης Οκτωβρίου 2019 που απεστάλησαν με email στις 2 Οκτωβρίου με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού θα θεωρηθούν εγκεκριμένα μιας και μέχρι 4 Οκτωβρίου δεν εκφράστηκαν αντιρρήσεις. να ξεκινήσουμε με το βραβείο Λουξ. 13 χρόνια μετά την δημιουργία του, το βραβείο ταινιών Λουξ εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο. Όλο και πιο σημαντικό μάλιστα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία βασίζεται και επικεντρώνεται σε ευρωπαϊκές αξίες και ευρωπαϊκά θέματα που στηρίζουν τις αρχές του ευρωπαϊκού έργου. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει επίσημα η ιστορική αυτή διαδικασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέσο Video On Demand και μέσω πακέτων DVD για τους ευρωβουλευτές. Επίσης ξεκινάει η διαδικασία ψηφοφορίας και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως πρεσβευτές για το βραβείο αυτό. Φέτος λοιπόν έχουμε τα εξής, ε, τις εξής ταινίες. Cold Case, Hammarskjöld του Mats Brügge. God exists. Her name is Petrunia. Tis Teona Strugar Mitevska. The Realm του Ροντρίγκο Sorogoyen. Οι τρεις ταινίες λοιπόν θα προκληθούν ε, στις Βρεξέλλες από 11 έως 22 Νοεμβρίου στο... στην αίθουσα Λούξε στο χώρο με Μεουνουντή και τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν από 24 Οκτωβρίου μέχρι 26 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ μέσα από την ιστοσελίδα www.luxprice.eu, κάθετος vote. Το, η γραμματεία για το βραβείο Lux μπορεί να σας υποδείξει πού μπορείτε να βρείτε το κάθε έργο. Και την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, θα απονεμηθεί το βραβείο τελικά στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια. Φυσικά το θέμα δεν είναι μόνο ποια ταινία θα, ποια θα κερδίσει. Το θέμα είναι να προβληθούν οι ταινίε όσο πιο πολύ γίνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη. Και γι' αυτό λοιπόν ε, τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν οργανώσει τις Lux Film Days, τις ημέρες ε, ταινιών το πρόγραμμα Simultaneous Screening, στο οποίο συνεργάζεται από κοινού με το δίκτυο Creative Europe Media και προβάλλεται σε σινεμά. 6, 7 και 8 Νοεμβρίου λοιπόν θα προβληθούν οι τρεις ταινίες σε 15 ευρωπαϊκές χώρες και στην Ισλανδία, τη Βόρειο Μακεδονία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Οι τρεις Συντελεστέ των ταινιών θα εμφανιστούν στις Βρυξέλλες ε, στην αίθουσα Μποζάρ και στις, ε, στους κινηματογράφους για να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση η οποία θα μεταβληθεί ζωντανά θα μεταδοθεί ζωντανά σε 35 κινηματογράφους. Οι συζητήσεις θα προβληθούν επίσης ε, ζωντανά στο Facebook και στην ιστοσελίδα του Άρτα. Επίσης ξεκίνησε η 8η έκδοση των Lux Film Days. Οι τρεις ταινίες Lux ε, θα προβληθούν πάνω από 200 φορές από τον Οκτώβριο στο Δεκέμβριο σε όλη την Ευρώπη και τα μέλη τα οποία θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση μπορούν είτε να αποτανθούν στη γραμματεία του βραβείου Lux είτε στο γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της κάθε χώρας. Και είναι όλο και πιο πολλοί αυτοί οι ευρωβουλευτέ που θέλουν να οργανώσουν προβολέ των ε, ταινιών του βραβείου Λούξ ε, στι περιφερειέ του. Και έχετε λοιπόν ένα εγχειρίδιο με διάφορε πρακτικέ ε, πληροφορίε για την οργάνωση μια τέτοια προβολή. Και έχετε ήδη λάβει επίση και ένα φυλάδιο για την φετινή έκδοση του βραβείου Λούξ, τον κατάλογο των τιμών σε ό,τι αφορά το βραβείο Lux και ένα DVD με τις τρεις ταινίες και 24 ε, υποτίτλους. Στα πλαίσια λοιπόν της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ταινιών έχουμε κάποιες θέσεις που περισσεύουν σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό, στην ε, Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για την αποδοση, απονομή των βραβείων στο Βερολίνο. Αλλά δεν έχουμε ωστόσο δικαίωμα για έξοδα ταξιδίου και παραμονής στο Βερολίνο. Το βραβείο λοιπόν ε, Λούξ ε, πάντα προβάλλεται και στα διεθνή φεστιβάλ και στο Βερολίνο, στις Κάνες και στην Βενετία. Και εδώ είναι σημαντικό να υπάρχει παρουσία μελών της Επιτροπής Πολιτισμού. Τα φεστιβάλ ε, είναι άλλωστε ιδανικές ε, περιστάσεις προκειμένου να ξεκινήσουμε διάλογο με διάφορες οργανώσεις, ενώσεις και εταίρους. Η παρουσία λοιπόν των Ευρωβουλευτών είναι πολύ ευκταία. Αν θέλετε λοιπόν, αποτανθείτε και πάλι στη γραμματεία του βραβείου Λουξ. Αγαπητοί συνάδελφοι, το βραβείο Λουξ δεν αποτελεί μόνο σημαντική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά έχει και μια εξαιρετική ευρωπαϊκή πολιτισμική υπεραξία. Η Επιτροπή μας λοιπόν θα πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα. Να συζητήσουμε λοιπόν και να συζητάμε τις ταινίε με τους συναδέλφους μας και να τους πείσουμε να πάνε να δουν τις ταινίε αυτές και να ψηφίσουν. Σας καλώ λοιπόν ως μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού να δραστηριοποιηθείτε πιο ενεργά για το βραβείο Λούξου. Θα συνεχίσουμε. Όπως τα ξέρετε, τα μέλη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης του προϋπολογισμού μπορούν να προτείνουν διάφορα πολιτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικά μέτρα μετά από πρώτο έλεγχο από πλευρά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα καλύτερα αυτά έργα ε, θα εγκριθούν από τις Επιτροπές και από την Ολομέλεια. Τα έργα που θα εγκριθούν θα εκτελεστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην τρέχουσα λοιπόν θητεία θα θέλαμε να εξετάσουμε πιο α, στενά την εκτέλεση των έργων αυτών και θα θέλαμε να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάζει τακτικά διάφορα τέτοια έργα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τέσσερα τέτοια έργα τα οποία θα μας παρουσιάσει η Γενική Διεύθυνση ΕΑ και η Γενική Διεύθυνση ΣΥΝΕΚΤΑ. Και θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν τους προσκεκλημένους μας από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Ingrid Ρίγκλερ, η οποία είναι Ματάρχησα στην Γενική Διεύθυνση ΕΑΚ και η οποία θα μας κάνει μια γενική εισαγωγή σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης των PPAs. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που καλέσατε την Κομισιόν για να σας παρουσιάσουμε ορισμένα πλειοτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ε, δράσεις τις ε, οποίες ε, εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή. Για να κάνουμε κάτι τέτοιο καλύτερα να ξεκινήσω με μια σύντομη εισαγωγή για το πώς αξιολογούμε αυτά τα σχέδια και αυτές τις δράσεις που παίρνουμε από το Κοινοβούλιο και ποια κριτήρια χρησιμοποιούμε. Καταρχήν θα ήθελα να δούμε τον ορισμό των προ, προπαρασκευαστικών δράσεων και των πιλωτικών σχεδίων σύμφωνα με τον χρηματοοικονομικό κανονισμό. Αυτά τα σχέδια και οι δράσεις ε, λειτουργούν χωρίς ε, νομική βάση και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Κομισιόν. Αυτές είναι οι βασικές ε, αρχές για την αξιολόγηση των σχεδίων και των δράσεων. Τα πιλωτικά σχέδια βρίσκονται λοιπόν εναντίον, ε, ε βρίσκονται εντός των ευρωπαϊκών ε, αρμοδιοτήτων και εκτός νομικής βάσης, ε, ενώ μαζί με τις προπαρασκευαστικές δράσεις ε, χρησιμεύουν για να προετοιμάσουμε καινούριε νομοθετικές προτάσεις. Να δούμε τις διάφορες κατηγορίες που διαθέτουμε. Έχουμε τέσσερις συγκεκριμένες κατηγορίες, A, B, C και D. Για να δούμε ποιες είναι. Καταρχήν, να πούμε ότι κατά την αξιολόγηση των προτάσεων που προέρχονται από, την, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιούμε νομικά, αυστηρά νομικά κριτήρια. Το οποίο σημαίνει ότι η κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί κάποια οποιαδήποτε πρόταση δεν έχει σχέση με την αξία του ίδιου του σχεδίου ή της δράσης. Για παράδειγμα, αν η πρότασή σας ενταχθεί στην κατηγορία C ή στην D, δεν σημαίνει ότι είναι κακή η πρόταση το περιεχόμενό της, ε, απλά εκεί πέφτει, εκεί εντάσσεται με βάση τα νομικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούμε. Ας τις δούμε λοιπόν αυτές τις κατηγορίες. Κατηγορία Α. Αυτά που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία σημαίνει ότι μπορούν να εφαρμοστούν ακριβώς όπως προτάθηκαν. Ακριβώς λέω όπως προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούν αυτές οι προτάσεις να καλυφθούν από υπάρχοντα προγράμματα. Δεν υφίσταται βέβαια νομική βάση. Θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτές οι προτάσεις εκτός νομικής βάσης. Και επίσης αυτές οι προτάσεις δεν μπορούν να ενταχθούν σε οποιοδήποτε τρέχον ισχύον πρόγραμμα. Δεύτερη κατηγορία, κατηγορία B. Είναι προτάσεις που θα μπορούσαν οι υποσυγκεκριμένες συνθήκες να εφαρμοστούν, αλλά το, η πρόταση, το σχέδιο θα πρέπει εν μέρη να αναδιαρθρωθεί, διότι εν μέρη μπορεί να καλύπτεται από υφιστάμενη νομική βάση ή από κάποιο ή κάποια πρόταση είναι υπερβολικά φιλόδοξη και δεν μπορεί να καλυφθεί με τον προϋπολογισμό που διαθέτουμε. Συνεπώς, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση που εμπίπτει στην κατηγορία B, θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Ενδεχομένω επίσης μπορεί η Κομισιόν να μην έχει αρκετέ πληροφορίε και να ζητά πληροφορίες ε, όταν εντάσσει σχέδια σε αυτήν την κατηγορία. Κατηγορία C. Αυτές οι προτάσεις καλύπτονται πλήρω από μία εφιστάμενη νομική βάση ή από κάποιο άλλο πιλωτικό σχέδιο ή προπαρασκευαστική δράση. Και πάλι επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για κακέ ιδέε, απλά λέω ότι είναι ιδέε, προτάσει που μπορούν να καλυφθούν από υφιστάμενα σχέδια. Και η τελευταία κατηγορία, η κατηγορία D, έχουμε για αυτήν την κατηγορία προτάσεις με, προβλήματα υλοποίησης, τυπικά προβλήματα ας πούμε, όπως για παράδειγμα γιατί η πρόταση αναφέρει συγκεκριμένο δικαιούχο, κάτι που αντιβαίνει με τον οικονομικό κανονισμό ή το θέμα διαφεύγει από τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες. Ε, για παράδειγμα, προβλέπει την ανάπτυξη ενός ε, εκπαιδευτικού προγράμματος ε, ή πρόκειται για κάποια καθαρά εθνικά προγράμματα, σχέδια εθνικής και μόνον εμβέλειας. Αυτά είναι τα κριτήριά μας σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση. Θα σταματήσω εδώ και πολύ ευχαριστώ θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα πιλωτικά προγράμματα, αν έχετε ερωτήσεις για κάποια δικά σας, κάποιες δικές σας προτάσεις, πολύ ευχαριστώ να σας να τις σημειώσουμε και να σας απαντήσουμε διμερώς, διότι έχουμε δεκάδες πιλωτικά σχέδια που τρέχουν αυτή τη στιγμή και φοβούμε ότι ε, δεν θα μπορούσα να απαντήσω λεπτομερώς ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις για το α ή το β πιλωτικό σχέδιο που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα πρότεινα Καταρχάς να ακούσουμε όλες τις παρουσιάσεις για όλα τα έργα και στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο για τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Σε κάθε ερώτηση να διευκρινίσετε σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας, για ποιο έργο δηλαδή. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στον κύριο Σόλτ Σοκολάη από την Γενική Διευθυνσία και Μονάδα Πολιτισμού θα μας μιλήσει για το έργο Music Moves Europe. Thank you very much. Uh, hello, good morning. Uh, I'm uh, briefly... Καλή σας ημέρα. Θα σας κάνω μία σύντομη παρουσίαση της προπαρασκευαστικής δράσης που ψηφίστηκε πρώτα το 2018 και από το Κοινοβούλιο και ε, χρηματοδοτήθηκε με 500.000 ευρώ ε, και μετά ε, με 3 εκατομμύρια ευρώ ε, και μάλιστα έχει ήδη προταθεί να συνεχιστεί τον επόμενο χρόνο. Πρόκειται για την πρόθεση της μουσικής ε, διαφορετικότητας ε, στην Ευρώπη. Πρόκειται για προπαρασκευαστική δράση η οποία θέλει να προωθήσει την πλέον κατάλληλη δράση η οποία θα υποστηρίξει πλήρως την μουσική ε, μέσω μελλοντικών υποστηρικτικών πολιτιστικών προγραμμάτων. Ε, καλωσορίζουμε την, καλοδεχόμαστε την ε, ιδέα αυτή, έστω και αν δεν εντάσσεται πλήρως στο πρόγραμμα Creative Europe, Δημοκρατική Δημιουργική Ευρώπη, γιατί προωθεί ε, πλην δύο στοιχείων ε, όλες τις τέχνες, ωστόσο η μουσική δεν αναφέρεται ε, ιδιαίτερα ή ξεχωριστά. Λόγω της ψηφιοποίησης στον τομέα της μουσικής όμως θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και οπωσδήποτε η μουσική να προστατευτεί. Πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα την αγορά γιατί δεν έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας πάρα πολλά στοιχεία και θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς που θα επιτρέψουν την καλύτερη επιτήρηση. Ταυτόχρονα να βελτιώσουμε την κινητικότητα των καλλιτεχνών μέσα από ε, διαδικασίες οι οποίες θα τους κάνουν και πιο ανθεκτικούς απέναντι στην αγορά. Τρίτο στοιχείο είναι να δοκιμάσουμε ε, διάφορα μοντέλα ε, διανομής έτσι ώστε εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, να κυκλοφορεί καλύτερη μουσική. Τέταρτο δε, ε, ε, θέλουμε να δούμε πώς είναι δυνατόν σε μια διαφοροποιημένη αγορά να προστατέψουμε το μπραντ. Είχαμε δύο μελέτες και δύο call for proposals. Ε, οι δύο αυτές αφορούν την, ε, τον έλεγχο ε, πρωτοποριακών προγραμμάτων για επιγραμμική και μη διανομή, έτσι ώστε να δούμε με ποιο τρόπο καλύτερα μπορούμε να φτάσουμε στο ακροατήριο. Όσον αφορά την κατάρτιση, ζητούμε βελτίωση της επαγγελματικής ας πούμε κατάρτισης ε, και εδώ δεν αναφερόμαστε στην καλλιτεχνική δημιουργία όσο ε, στις ε, ικανότητες τις επιχειρηματικές. Είχαμε όπως σας είπα και δύο διαδικασίες προσφορών και δύο διαδικασίες μελετών, μελέτη για την αγορά αφενός και μελέτη για το παρατηρητήριο εφετερού. Τα projects έχουν ήδη ε, ξεκινήσει, ε, θα ολοκληρωθούν περί τον Μάρτιο του 2020. Όσον αφορά τώρα ε, για το θέμα της διανομής, οργανώνουμε μια συνάντηση διαλόγου τον μήνα Δεκέμβριο, έτσι ώστε να κατανοήσουν οι δύο πλευρές η μία την άλλη και ε, αυτό θα ολοκληρωθεί επίσης ε, και τον Μάρτιο. Όσον αφορά τις μελέτες, περιμένουμε ε, τελικά αποτελέσματα περί τα τέλη τρέχοντος έτους και οπωσδήποτε θα προβλέψουμε και το, την απαραίτητη παρακολούθηση follow-up σύμφωνα με τα όσα θα αναφέρονται σε τις μελέτες αυτές. Το 18, μετά το 18 λοιπόν διπλασιάστηκε ο προπολογισμό και αποφασίσαμε να διευρύνουμε και το, τα προγράμματα αυτά. Συνεχίζουμε με την κατάρτιση γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για τέτοια κατάρτιση. Και ε, μετά τα αποτελέσματα της ε, ε, στρατηγικής ε, των εμπειρογνωμόνων θα προχωρήσουμε και στην ολοκλήρωση προγραμμάτων βάσει των ευρημάτων αυτής της μελέτης. Όσον αφορά την διανομή, αποφασίσαμε να, να ασχοληθούμε με μικρά κλαμπ, μικρές αίθουσες οι οποίες αποτελούν κατά κάποιο τρόπο την, τις με θερμοκοιτίδες πούμε ε, όπου αναπτύσσονται νέες τάσεις. Αποφασίσαμε να κάνουμε και μια νέα προκήρυξη για τη συνδημιουργία έτσι ώστε να ε, βάλουμε, να δώσουμε τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να συνεργαστούν και να ελέγξουν ε, τα αποτελέσματα της συνεργασίας όσον αφορά την καλλιτεχνική κατάρτιση και την καλλιτεχνική παραγωγή. Ήδη ε, ετοιμάζουμε και ένα εργαστήριο σχετικά με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι μουσικοί στην κατάρτισή τους αλλά και στην επαγγελματική τους ε, πορεία. Τα αποτελέσματα σύντομα θα δημοσιευτούν. Και να σας πω γενικότερα ότι στόχος ε, είναι να ελέγξουμε νέες ιδέες. Συνεργαζόμαστε βεβαίως και με όλες τις χώρες μέλη στο Συμβούλιο. Συζητούμε τις ε, ανάγκες ε, του ε, μουσικού τομέα. Βεβαίως μελετούμε και όλες τις παρενέργειες κατά κάποιο τρόπο ή επιρροές των θεμάτων πνευματικής διανοητικής ιδιοκτησίας. Εμείς ελέγχουμε και αμοιβαία τα ευρήματα με άλλους τομείς ε, έτσι ώστε ε, να έχουμε μια συνολική ευρωπαϊκή τομεακή προσέγγιση όσον αφορά τη μουσική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Μαρίζα Φερνάντα Αστεμπάνο η οποία είναι από τη Γενική Διεύθυνση ΑΚΑ για να μας παρουσιάσει το έργο ε, αθλητισμός ως εργαλείο για την ε, ένταξη και την κοινωνική συμπερίληψη των προσφύγων. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω για πράγματι για το σχέδιο αυτό που έχει σχέση με τον αθλητισμό ως εργαλείο για την ένταξη και κοινωνική ε, ενσωμάτωση των μεταναστών. Ε, είναι βασική προτεραιότητα στον τομέα του αθλητισμού. Έχουμε το πρόγραμμα Erasmus Plus για αυτήν και για άλλες προτεραιότητες. Ο αθλητισμός μπορεί να χρησιμεύσει σε μεγάλο βαθμό στην ένταξη των μεταναστών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά σχέδια σε όλη την Ευρώπη, σε τοπικό επίπεδο, σε επιφυλακό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για να βελτιώσουν την ένταξη των μεταναστών σε όλη την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, μέσω του Erasmus Plus υπάρχει μια ανάγκη η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί. Γιατί το Erasmus Plus δεν αναφέρει τίποτα συγκεκριμένο για την ένταξη των μεταναστών στην νομική του βάση. Δεδομένω όμω τη ε, απόλυτη σημασία αυτή τη προτεραιότητα τη ένταξη των μεταναστών, θεωρήσαμε ότι αυτό είναι ένα κενό που θα έπρεπε να καλυφθεί με τέτοιου είδους προπαρασκευαστικές δράσεις και πιλωτικά προγράμματα. Ένας από τους ε, στόχους αυτής της ε, δράσης και του σχεδίου είναι να βοηθήσουμε τις διάφορες οργανώσεις να συνεργαστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν βέλτιστες ε, πρακτικές ε, και να εντοπίσουν τον καλύτερο τρόπο ένταξης των μεταναστών μέσω του αθλητισμού. Μέχρι το 2019 ε, χρηματοδοτήσαμε 54 σχέδια με μέγιστο προϋπολογισμό 60.000 ευρώ με βασικό στόχο τις ε, τοπικές οργανώσεις, αθλητικές οργανώσεις, ε, αθλητικά ιδρύματα και ομοσπονδίες. Βλέπετε ότι ο προπολογισμό ε, αυξάνεται. Το 2016 0,6 εκατομμύρια ευρώ με 53 αιτήσει και 11 επιλεγμένα σχέδια. Το 2017 1 εκατομμύριο ευρώ, 111 αιτήσει, 19 επιλεχθέντα σχέδια. Το 2018 1,4 εκατομμύρια ευρώ, 96 αιτήσει είχαν ληφθεί το 2018 και είχαμε επιλέξει 24 σχέδια. Φέτο έχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο προπολογισμό, πολύ μεγαλύτερο 3 εκατομμύρια ευρώ, με δύο προσκλήσει εκδήλωση ενδιαφέροντο. Ε, η πρώτη έχει σχέση με τη συνέχεια παλιότερων προγραμμάτων, η δεύτερη για αθλητικές δραστηριότητες, για πιο μακροχρόνια σχέδια για παράδειγμα προετοιμασία και εκπαίδευση ε, προπονητών και προσωπικού που θα δουλέψει στην ένταξη και επίσης ε, δικτύωση και διάδοση των αποτελεσμάτων. Θέλουμε δηλαδή να συνδέσουμε τα αποτελέσματα των σχεδίων σε διάφορες χώρες. Έχουμε λάβει 70, λάβαμε 70 αιτήσει και επιλέξαμε 11 προγράμματα. Αυτή είναι αυτός είναι ο κατάλογος των 11 αυτών προγραμμάτων που επιλέξαμε. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα αυτά. Βλέπετε ότι έχουμε εδώ σχέδια από διάφορα κράτη-μέλη. Και μια ποικιλία οργανώσεων. Για παράδειγμα, το πρώτο, Deutsche Olympischer Sportbund από τη Γερμανία. Έχετε μια μη κυβερνητική οργάνωση από την Ιταλία. Ε, το, ε, το αθλητικό κλαμπ ε, η αθλητική λασκή εκβόντω από την Κροατία. Έχετε την, βλέπετε την πόλη της Μούρθια από την Ισπανία την ε, Ποδοσφαιρική Ένωση Μάλτας, το Βέλγιο, το ποδοσφαιρική ομάδα του Κράινεμ, μια μικρή ποδοσφαιρική ομάδα στο Βέλγιο, η, την μη κυβερνητική οργάνωση Play International της Γαλλίας και μια μεγάλη μη κυβερνητική οργάνωση της Δανίας. Βλέπετε έχουμε μια μεγάλη ποικιλία ε, φορέων οι οποίοι επιλέχθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Έστεμπαν και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Λουτσία Ρεκάλτα η οποία είναι ε, επικεφαλής στη μέσων ενημέρωσης στη Γενική Διευθύνση Connect η οποία θα μας ε, δώσει μία παρουσίαση για το έργο για τον υποτετλισμό Ευρωπαϊκού ελληνικής ε, πολιτισμικής τηλεόρασης και περιεχομένων σε όλη την Ευρώπη. Thank you very much, uh, Chair, and thanks for giving me the opportunity to present to you. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω αυτό το pilot, το πιλωτικό πρόγραμμα ε, και την προπαρασκευαστική δράση σχετικά με τον υποτιτλισμό. Στόχος ε, αυτής της προπαρασκευαστικής δράσης και τη, για τον υποτιτλισμό είναι να προσπαθήσει να δημιουργήσει και χρησιμοποιήσει καινοτόμες στρατηγικές ε, όσον αφορά τον υποτιτλισμό ε, ε, πολλών ευρωπαϊκών πολιτιστικών προγραμμάτων κύριο κριτήριο επί τη βάση του οποίου ξεκινήσαμε τον ε, διαγωνισμό ήταν ε, η ε, προσφορά τουλάχιστον 300 ώρων υποτιτλισμένου πολιτιστικού περιεχομένου. αυτή τη στιγμή το Arte, Arte Europe και το Europa μέσω του VPRO χρησιμοποιούν συμμετέχουν στη δράση αυτή. Ε, η πρώτη πιλωτική φάση ξεκίνησε το 2015 και τότε ο μόνος ε, ε, We got two proposals in... Δικαιούχος ήταν το Άρτε, μετά το 2016 προσθέθηκε το VPRO. Είχαμε ξανά μετά δύο υποψηφίους το 17, ενώ το 18 μονάχα έναν υποψήφιο ε, και το 19 είχαμε κύριο δικαιούχο τη VPRO από το 19 ε, το ΑΡΤΕ θα λαμβάνει χρηματοδότηση ε, όσον αφορά τον υποτιτλισμό από μια νέα δράση. Γι' αυτό ακριβώς έχει αφαιρεθεί ε, το ΑΡΤΕ από αυτό το συγκεκριμένο πιλωτικό πρόγραμμα και νομίζω ότι αυτό αποτελεί και απόδειξη πως ένα πρόγραμμα όπως το Media μπορεί να προωθήσει τέτοιου είδους ε, δράσεις. Ε, το VPRO έχει ε, δώσει υποτιτλισμό σε αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά μέσω του καναλιού YouTube και έχει αυξήσει την, την παρακολούθησή του. Να σας πω δύο λόγια και για την εμπειρία της Άρτε. Η Άρτε βασίστηκε ε, στην ε, γνώση και την τεχνογνωσία που είχε ήδη στα γερμανικά και τα ε, γαλλικά. Ε, και μέσω της δράσης αυτής ε, το, και το Κοινοβούλιο διεύρυνε, ε, διεύρυνε την προσφορά στα Ισπανικά και μετά Πολωνικά και Ιταλικά. Είναι πολύ μεγάλη η προστιθέμενη αξία αυτού του προγράμματος. Είναι αδιαμφισβήτητη δε με την έννοια ότι μέσω αυτής της διάταξης του πολιτιστικού περιεχομένου σε έξι ευρωπαϊκές γλώσσες 70% των Ευρωπαίων πολιτών έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο στη δικιά τους γλώσσα. Αυτό το περιεχόμενο ε, δεν είναι διαθέσιμο μόνο στην Ευρώπη, αλλά ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ξέρουμε ας πούμε ότι στις Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για κάποιο από το περιεχόμενο που προβάλλει το Άρτε μέσω της αγγλικής εκδοχής. Ε, θεωρήσαμε ότι αυτό το project ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο και θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να μοιραστούμε τα αποτελέσματα με όλη την ε, Επιτροπή. Γι' αυτό ε, ξεκινήσαμε μια σειρά συζητήσεων και συναντήσεων ε, ε, διανομής ή προώθησης αν θέλετε ε, πρώτα απ' όλα 19 ε, και Απριλίου του 2018 στις ε, Βρυξέλλες ε, και σε συνεργασία με την DG Connect στη 31 Μαΐου του 2018 πάλι στις Βρυξέλλες έτσι ώστε να προωθήσουμε τον υποτιτλισμό και να είναι ευρύτερα διαθέσιμος. Τι διδαχτήκαμε. Πρώτα απ' όλα ότι ο υποτιτλισμός μπορεί να έχει πάρα πολύ θετικό, θετική επίπτωση στην κυκλοφορία ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσης, ε, ε, είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μοντέλο με την έννοια ότι ε, προωθείται ο υποτιτλισμός από την ε, εταιρεία η οποία έχει λάβει χρηματοδότηση ε, και η οποία συμπληρωματικά χρηματοδοτεί και εκείνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να αναπτύξουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική επικοινωνίας η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τη διαφορετικότητα, τις ιδιαιτερότητες των γλωσσών και των περιφερειών και με τον τρόπο αυτό να ε, είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε στην ανάγκη ε, ε, αποτελεσματικής προσφοράς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα για την τελευταία παρουσίαση. Μπορώνα Βόλτον θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα Media Literacy for All. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω πολύ που με επιτρέψετε να παρουσιάσω το πορίσμα, τα πορίσματα του Media Literacy for All. Αυτό ήταν λοιπόν ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε το 2016 και σκοπός μας ήταν να βελτιώσουμε τον αλφαβητισμό σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωση για όλους. Αυτό πάντα αποτέλεσε σημαντικό θέμα για τις ομάδες, ε, τις μειονεκτικές, τις ε, ομάδες ε, των ατόμων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας. Σκοπός, λοιπόν, ήταν να βελτιώσουμε την ικανότητα των πολιτών να αξιολογούν το περιεχόμενο που λαμβάνουν μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και νομίζω ότι το θέμα του αλφαβητισμού στα μέσα ενημέρωση είναι ένα θέμα το οποίο αποτελεί κλειδί για πολλού από εμά. Από το 2016 έως σήμερα λοιπόν το θέμα αυτό και το έργο αυτό μας επέτρεψε να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις αλλαγές που ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης. Έχουμε λάβει λοιπόν υπόψη αυτή την τεράστια αλλαγή η οποία έχει λάβει χώρα και το εργαλείο είναι πάρα πολύ ευέλικτο σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που διαδραματίζονται στα μέσα ενημέρωση. Ένα σημαντικό θέμα ήταν ε, η αλλαγή του πώς αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης πλέον οι πολίτες. Αρχικά λοιπόν, κοιτάξαμε το θέμα της εκπαίδευσης πώς ε, ε, συμπεριφερόμαστε σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο στα μέσα ενημέρωση και σκεφτόμαστε πιο πολύ τον τελευταίο καιρό το ρόλο των ίδιων των πολιτών. Όταν εμφανίζονται στο διαδίκτυο, online, πώς κάνουμε like, πώς ε, μοιραζόμαστε περιεχόμενο, ιδιαίτερος σε ό,τι αφορά τα, τις ειδήσει. Θεωρούμε ότι όλοι μας πλέον είμαστε τμήμα του περιβάλλοντος των μέσων ενημέρωσης, γιατί συχνά μοιραζόμαστε με άλλους ιστορίες και συχνά ιστορίες οι οποίες ενδεχομένως να είναι παραπλανητικές. Ένα από τα άλλα σημαντικά στοιχεία ήταν να κινηθούμε από έργα τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε νέους και να συνδεθούμε και να συσχετιστούμε και με άλλους μεγαλύτερους ε, σε ηλικία πολίτες. Γιατί προφανώς ε, οι νέοι είναι πιο πολύ σε θέση να προσαρμοστούν στο ψηφιακό περιβάλλον. Αλλά συχνά οι πιο ηλικιωμένοι είναι αυτοί που ζορίζονται να καταλάβουν ποιε είναι οι συνέπειε των δράσεών τους online και να κατανοήσουν κατά πόσον οι πληροφορίε που λαμβάνουν είναι αξιόπιστες. Άρα, συνολικά, από τότε που προγραμματίσαμε το έργο, ξεκινήσαμε με ένα πολύ μικρό προϋπολογισμό. Έχουμε 250.000 λοιπόν ευρώ. Έχουμε χρηματοδοτήσει δύο έργα. 125.000 έκαστο. Το δεύτερο έτος λάβαμε 500.000 και καταφέραμε να χρηματοδοτήσουμε άλλα τέσσερα έργα. Το τέταρτο έτος, το τρίτο έτος τα ίδια, 500.000 και τέσσερα έργα. Σας είπα, ε, ότι επικεντρωνόμαστε πέρα από τα παραδοσιακά προγράμματα εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης. Το 2017 χρηματοδοτήσαμε έργα όπου εξετάσαμε τον αντίκτυπο των πληροφοριών που παρέχονται online στα μέσα ενημέρωσης, το πώς παρουσιάζονται οι γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης και κυρίως ό,τι αφορά την υγεία των γυναικών. Επίσης, ε, κοιτάζουμε το θέμα των μέσων ενημέρωσης ε, από πλευράς ε, της δημοσιογραφίας, σε ό,τι αφορά φοιτητές δημοσιογραφίας. Επίσης, υποστηρίξαμε και χρηματοδοτήσαμε έργα για να υποστηρίξουμε τους fact-checkers, αυτούς που ελέγχουν κατά πόσον στέκουν τα όσα αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης. και θεωρούμε ότι αυτά θα μας δώσουν σημαντική προπαρασκευαστική αξία σε ό,τι αφορά το θέμα του γραμματισμού της παιδείας στα μέσα ενημέρωσης ε, για την περίοδο του 2020. Και τέλος, θα ήθελα να σας ζητήσω να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αναμειχθείτε κι εσείς ε, στην εβδομάδα παιδείας στα μέσα ενημέρωσης. Ε, Μαρτίο και Απρίλιο θα λάβει η χώρα του 2020. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, Media Literacy, θα διοργανώσουμε μια, ένα συνεδρίο στο Ζάγκρεπ για θέματα τα οποία μας απασχολούν ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Warden, για την παρουσίασή σας. Αγαπητοί συνάδελφοι. ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα με τον γύρο των ερωταπαντήσεων. Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας. Παρακαλώ να μας πείτε σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας και θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία ping-pong για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Θα ακούμε δηλαδή ερώτηση-απάντηση. Να ξεκινήσουμε με τον πρώτο βουλευτή. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση για την κυρία Ρίγκλερ. Πραγματικά να σας πω ότι απογοητεύτηκα από αυτά που άκουσα. Τα κριτήρια δεν έχουν αξιοπιστία και νομίζω ότι αυτό που είναι προφανές είναι ότι έχετε ε, ένα πρόγραμμα, μία ατζέντα βάσει των οποίων επιλέγετε τα προγράμματα τα οποία μπορούν να κουμπώσουν μέσα σε αυτό το, ε, το πρόγραμμα, σε αυτή την ατζέντα. Ε, Ας πούμε, ε, απορρίψατε κάποια πιλωτικά προγράμματα επί τη βάση της εσφαλμένης, ας πούμε, δημοσιονομικής γραμμής ε, ή ε, είπατε ότι είναι D ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο... Ustedes decían que no entraba en su ámbito de competencia proponer un acto interinstitucional con el Consejo y con el Parlamento Europeo. Ε, γιατί ε, δεν εντάσσεται στην 70η ε, επέτειο της, από τη γέννηση του Σούμαν. Επίσης είπατε ότι διευρύνεται την ε, ε, δικαιοδοσία της Κομισιόν να προβάλλει ε, κάποιο βιογραφικό ας πούμε ή κάποια, κάποιο κουρίκουλουμ για, την, για το ευρωπαϊκό έτος αλλά δεν είναι δυνατόν να μας παίρνετε για χαζούς δεν είναι δυνατόν να μας κοροϊδεύετε με αυτόν τον τρόπο. Διαφορετικά, εάν έχετε πραγματικά ε, γνωμοδότηση της ε, ε, νομικής υπηρεσίας που μπορείτε να, βάλετε και τέτοια στοιχεία και να βάλετε εσείς υποδείξεις να κάνετε στα κράτη-μέλη, να μας πείτε, να μας τη δείξετε αυτή την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Yes, thank you for your question. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας, λέει η κυρία Ρίγκλερ. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να επαναλάβω αυτό που είπα και πριν, δηλαδή ότι δεν κρίνουμε ε, τα προγράμματα ε, ε, βάση της αξίας τους, αλλά και βάση κυρίως των νομικών προϋποθέσεων και απαιτήσεων. Είναι γεγονός ότι πρόκειται για μία νομική ε, αξιολόγηση για το κατά πόσον μπορεί να ε, έχει δικαίωμα και πρόσβαση σε χρηματοδότηση ένα τέτοιο πιλωτικό πρόγραμμα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να ενταχθεί στο πιλωτικό σχήμα όσον αφορά τα όσα αναφέρατε σχετικά με το D, είναι γεγονός ότι πάντα βάσει νομικής ε, ε, γνωμοδότησης, εάν θεωρήσουμε ότι κάποια ε, προγράμματα δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν, τότε θα πρέπει να τα βάλουμε στην κατηγορία D. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε ε, δεν κατάλαβα πολύ καλά το σχόλιο σας για το κουρίκουλουμ, αλλά πάντως μπορώ να σας πω ότι είναι γεγονός ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένες ε, δικαιοδοσίες όσον αφορά την εκπαίδευση. Ναι, αλλά υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο, στην πρόταση ενός κουρίκουλουμ και στην επιβολή ενός κουρίκουλουμ Αναφέρεται γραπτά ότι ε, τα, μέλη, τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία τα οποία είναι υπεύθυνα για, την, ε, ε, για το πρόγραμμα σπουδών, για το κουρίκουλουμ και το περιεχόμενό τους. Επομένως, δεν είναι δυνατόν εμείς να κινηθούμε διαφορετικά. Τα κράτη αποφασίζουν για τα προγράμματα σπουδών και το τι θα διδάσκεται στα σχολεία. Ο πρόεδρο, υπάρχει πάντα δυνατότητα να τα γραπτά τα ερωτήματά σα, γιατί δεν είναι δίκαιο να στερήσουμε το χρόνο των άλλων συναδέλφων. Μακρηγορώντα υπερβολικά. Η επόμενη ομιλητρία. Bunting? <laughs> Um, Συγγνώμη, το μικρόφωνο δεν μπορούσα να βρω. Και εγώ έχω μια ερώτηση να κάνω για, τα προτινόμενα έργα. Δεν ε, κρίνω εγώ αν ε, σωστά εγκρίνονται ή όχι. Αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι ότι και τα δύο έργα έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση στην επιστήμη, για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και για την προώθηση της εκπαίδευσης σε θέματα επιστημονικά για τα κορίτσια η επιστήμη και η μηχανική θεωρώ ότι αποτελούν ε, θεμελιώδη τμήμα τη πολιτισμού στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να τα βάλουμε σε μια γωνία σκονισμένη της επιστήμης πέρα από το πεδίο ε, της εντολής μας. Αλλά ανησυχώ γιατί και τα δύο προγράμματα καλύπτονται ήδη από άλλα προγράμματα χρηματοδότησης και αυτό τι σημαίνει συγκεκριμένα ότι πολύ απλά δεν υπάρχει νόημα Όποιος ε, και να προτείνει εδώ στην αίθουσα αυτή κάτι για να κάνει για την ε, επιστήμη. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε θα μας πούνε ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα επιστημονικό και να θέσουμε ως υποψήφιο πρόγραμμα θα καλύπτει την τον ορίζοντα ή από το Εράσμος. Ε, δεν πιστεύετε ότι κάποια προγράμματα έχουν να κάνουν με πιο εκπαιδευτικά ζητήματα τα οποία προέρχονται από το Εράσμους ή από τα υπόλοιπα προγράμματα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που δεν εμπίπτει στα δύο προγράμματα αυτά. Δεν μπορούμε να φανταστούμε κάτι παραπάνω. Yes, thank you for uh, question. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή και καταλαβαίνω Καταλαβαίνω απόλυτα τα πιλωτικά αυτά προγράμματα και προπροσκευαστικές αδράσεις που προτείνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά τα προγράμματα. Συγγνώμη, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να πει ότι κοιτάξτε εδώ βάζουμε κακό βαθμό γιατί καλύπτονται από τα άλλα προγράμματα. Αυτό όμως αποτελεί το νομικό ορισμό των πλητικών προγραμμάτων όπως ορίζεται στον χρηματοοικονομικό κανονισμό και αυτό υπό το τρέχον σύστημα, στους τρέχοντες κανόνες δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Τα έργα εκπαίδευσης, επιστημονικής εκπαίδευσης ε, θα μπορούσαν να ε, υποστηρίξουν ε, κάποια ένωση, κάποια οργάνωση πίσω από το έργο και να ζητηθεί χρηματοδότηση του έργου. Δεν σημαίνει δηλαδή το γεγονός ότι το έργο αυτό μπαίνει στην κατηγορία C. Αυτό το έργο δεν θα υλοποιηθεί, γιατί μπορεί να προκύψει ως πρόγραμμα το οποίο θα προταθεί από κάτω προς τα πάνω. Έτσι λειτουργούν τα προγράμματά μας. Μάλιστα, για να επιβεβαιώσω λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος εδώ στην αίθουσα να προτείνει κανείς κανένα πρόγραμμα για την εκπαίδευση την επιστημονική. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ ακραίο όπως το υποστηρίζετε. Αυτό προφανώς και εξαρτάται από το κάθε πρόγραμμα, από το κάθε έργο. Αυτό που έχω να σας προτείνω, αν έχετε εσείς ή κάποιος συνάδελφό σας μια ιδέα για ένα έργο και αμφιβάλλετε κατά πόσον καλύπτεται από την νομική μας βάση, να μας το πείτε, να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας και ανεπίσημα για να δούμε κατά πόσον καλύπτεται, κατά πόσον θα μπορούσε να μπει τμήμα του στην κατηγορία Β, για παράδειγμα, ενδεχομένω να μην καλύπτεται όλο το πρόγραμμα, αλλά κάποιο τμήμα αυτού. Ο πρόεδρο. Η κυρία Σόιτροβα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα προσεκτικά τα όσα ελέγχθησαν και η δική μας εμπειρία, πρέπει να πω, σε σχέση με τα πιλωτικά σχέδια είναι αρκετά θετική. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε το πώς σκέφτεται η Κομισιόν, ποιο σύστημα ακολουθεί. Για αυτά τα τέσσερα σχέδια τα οποία μας παρουσιάστηκαν, πρόκειται για προτάσεις οι οποίες συμπληρώνουν υφιστάμενα προγράμματα, τα οποία όμως δεν μπορούσαν να χρηματοδοθούν μέσω υφιστάμενων προγραμμάτων. Η επιστημονική κατάρτιση με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, οπότε θα μπορούσε να συμπληρώσει το Erasmus, το Erasmus Plus ή το Creative Europe, αν δεν, μπορεί να, αν δεν μπορούν να χρηματοδοθούν από το Erasmus Plus. Επίσης, η ένταξη των μεταναστών. Αν ένας φορέας ή μια πόλη αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα ενσωμάτωσης μεταναστών, ή κάποιων συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι νέοι, χρειάζεται να βοηθηθεί αυτή η πόλη ή αυτός ο φορέας. Όμως είναι δύσκολο να συμμετάσχει σε τέτοια σχέδια. ειναι έπρεπε να διευκολυνθούν Θα ήθελα να μου πείτε ποια ακριβώς, ε, ποιοι τύποι προγραμμάτων έχουν απορριφθεί και ποιοι έχουν γίνει δεκτοί. Ευχαριστώ κύριε Σόιτροβα. Νομίζω ότι αναφέρει την κυρία Στέβαν, έτσι δεν είναι η ερώτησή σας ε, αφορά την κυρία Στέβαν, φαντάζομαι. Yes, uh, thank you. Uh, Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ε, μία από τις προσκλήσεις εκδήλωση ενδιαφέροντος του Erasmus Plus όπως είπα και προηγουμένως, είναι για σχέδια τα οποία προωθούν την ενσωμάτωση ε, ομάδων του πληθυσμού. Εκεί δεν αναφέρεται ακριβώς ε, η ενσωμάτωση των προσφύγων. Ε, το προσφυγικό προέκυψε αργότερα και θα πρέπει να προβλέψουμε και τη δική τους ένταξη. Ο αθλητισμός είναι ένα καλό εργαλείο. Είναι πολύ εύκολο να διοργανώσουμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα με μια μπάλα μεταξύ δύο ομάδων που δεν χρειάζεται καν να έχουν κοινή γλώσσα. Μπορούμε να τους ε, βοηθήσουμε ταυτόχρονα και να μάθουν μια καινούργια γλώσσα και να βελτιώσουν τα προσόντα τους, ταυτόχρονα να καταρτήσουμε προπονητέ κλπ. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό τρόπο ένταξη. Θα είδατε την ε, παρουσίασή μου το πώς αυξάνεται κάθε χρόνο ο αριθμός των προτάσεων, ακριβώς γιατί είναι πολύ δημοφιλές ε, αυτό το εργαλείο. Λαμβάνοντας αυτές τις αιτήσει τις αξιολογούμε. Υπάρχει μια επιτροπή αξιολόγησης και κάθε πρόταση αξιολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τέσσερα κριτήρια τα οποία έχουμε. Μερικές φορές είναι δύσκολο να απορρίψουμε σχέδια γιατί πολλά σχέδια είναι ψηλής ποιότητας. Δυστυχώς όμως μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μόνο ένα συγκεκριμένο αριθμό σχεδίων εξαιτία του περιορισμένου προπολισμού που διαθέτουμε. Και χρειάζεται να βαθμολογήσουμε κατά κάποιο τρόπο τα σχέδια, αναγκαστικά. Θα θέλαμε να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε περισσότερα. Αλλά δυστυχώ περιοριζόμαστε από τον προπολογισμό μα. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σα. Äh, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Εστεμπάν. Η κυρία Κάμερφελτ, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι η παρουσίαση των προγραμμάτων, που, των projects που μόλις ακούσαμε, αποδεικνύει ότι είναι καλό ε, να γίνονται προσπάθειες στην προπαρασκευαστική φάση ε, και να, για να ξέρουμε αν τα προγράμματα αυτά μπορούν να ενταχθούν στα γενικά προγράμματα. Πρόκειται για πολύ καλά παραδείγματα, αυτά δηλαδή που αναφέρθηκαν και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί καλά και στο μέλλον η διαδικασία. Η επιλογή των πιλωτικών προγραμμάτων είναι πάντα δύσκολη, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια ε, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η επιλογή. Τώρα, κάποιοι συνάδελφοι δεν καταλαβαίνουν γιατί απορρίπτονται κάποια προγράμματα. Ε, νομίζω ότι και πάνω σε αυτό πρέπει να γίνει δουλειά. Θα πρέπει να ε, υπάρχει δυνατότητα εξήγησης γιατί ένα ε, project μπορεί να βρεθεί στην κατηγορία C ή ακόμα και στην κατηγορία D. Πάντως, σας ευχαριστούμε που μας προτείνετε να ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας. Ε, οποτεδήποτε πιστεύουμε ότι ένα εξαιρετικό project που ε, θα άξιζε να είναι πιλωτικό πρόγραμμα, να ε, το συζητήσουμε μαζί σας. Τώρα, η προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία είναι επίσης μια σημαντική αξία, ένα σημαντικό στοιχείο. Πολύ συχνά τα projects έχουν εθνική, ακόμα και περιφερειακή μονάχα ισχύ ή αξία. Πώς μπορεί να δοθεί λοιπόν αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση. Μιλήσατε επίσης ε, για ενσωμάτωση, πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και αυτό μέσω του αθλητισμού είναι γεγονός ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό συγκολητικό στοιχείο όχι μόνο για τους ε, πρόσφυγες αλλά και για τους ε, πολίτες γενικά. Κυρία Ρίγκλερ θέλετε να απαντήσετε παρακαλώ και μετά η κυρία Εστέμπαν. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι, βεβαίω, όταν αξιολογούμε τα, τα πιλωτικά προγράμματα πρέπει να ακολουθούμε μία συγκεκριμένη λογική ε, και να υπάρχει αυτή η συνεκτική, ας πούμε, λογική αντιμετώπιση ε, ε, για όλα τα προγράμματα, έστω και αν υπάρχουν πολλά αξιόλογα προγράμματα. Ίσως ναι, να πρέπει να εξηγήσουμε λίγο περισσότερο ευρύτερα γιατί ε, κάποιο πιλωτικό πρόγραμμα μπήκε σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Να δοθούν ε, ε, πιο ισχυρά επιχειρήματα έτσι ώστε όλοι να κατανοήσουν ότι μέσω των επιχειρημάτων ε, διαφαίνεται η σωστή αντιμετώπιση με την έννοια ότι το πιλωτικό πρόγραμμα δεν αντικατόπτριζε αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε και τα έτσι ώστε να μπει στην ε, κατηγορία Α. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, εγώ αναφέρθηκα προηγουμένως ε, σε δικτύωση και σε πρόθεση, networking and dissemination. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις ε, από τις πολύ μικρές αθλητικές οργανώσεις μέχρι τις πολύ μεγάλες που μπορεί να έχουν συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να διαλέξουμε τις πιο καλές ε, αιτήσει καλές όσον αφορά την δικτύωση και όσον αφορά την δυνατότητα να διατηρηθούν διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων projects. Δημιουργείται λοιπόν αυτή η κοινότητα χρόνο με το χρόνο και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να μιλάμε ε, για μια κοινότητα ενσωμάτωσης μέσω του αθλητισμού με γενικούς όρους, ε, όντως όχι μόνο για τους πρόσφυγες. Ε, κοιτάξτε, ε, ε, ένα πράγμα είναι το να παίξει κανείς σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, ένα δεύτερο πιο περίπλοκο είναι να ενταχθεί πραγματικά στην κοινωνία. Ωστόσο, και ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει μια γλώσσα επικοινωνίας Ξέρουμε ότι έχουμε ας πούμε ένα πρόγραμμα στο Κράινεμ στις Βρυξέλλες ε, για, ε, μη, ε, για συνόδευτα ανήλικα παιδιά. Εκεί γίνεται μια προσπάθεια και γλωσσική, δηλαδή βοήθεια στα μαθήματα, έτσι ώστε σιγά σιγά να αποκτήσουν και κάποιες κάποια προσόντα, κάποιες ε, εργασιακές ε, ικανότητες, δηλαδή συνεργασία ανάμεσα ε, σε προπονητές και δασκάλους. Και πραγματικά μιλάμε για προγράμματα πολύ ποιοτικά και ιδιαίτερα αξιόλογα. Frau Jembu, liebe Salima, du hast das Wort. Η Σαλίμα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ε, μία ερώτηση στην κυρία Εστεμπάν ε, σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης. Ε, όντως, ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει όχημα που θα οδηγήσει στην ενσωμάτωση, γιατί μεταφέρει ακριβώς ευρωπαϊκές αξίες, πολιτιστικές αξίες. Μπορείτε να μας πείτε, εάν σε αυτές τις οργανώσεις, σε αυτά τα project όλα, ποιο είναι το τμήμα ε, των ε, Ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή όχι μη προσφύγων. Υπάρχει ε, κοινωνική ανάμιξη όσον αφορά τη σύνθεση αυτών που ακολουθούν και συμμετέχουν. Αναφέρεστε πολύ συχνά στο ποδόσφαιρο. υπάρχει όμως κάτι άλλο, δηλαδή οι γυναίκες έχουν κάποια παρουσία και ποια είναι αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Γενμπού ήταν η ομιλήτρια. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γενμπού για την ερώτησή σας. Αν κατάλαβα καλά, η πρώτη σας ερώτηση ε, αφορά το κατά πόσον ε, συμμετέχουν μη πρόσφυγες και πόσοι είναι αυτοί. Το project ε, μέσω αυτής της πρόσκλησης ε, ενδιαφέροντος εμείς θελήσαμε να προωθήσουμε ε, την ε, ενσωμάτωση των προσφύγων στα πλαίσια του ευρύτερου Erasmus Plus ναι υπάρχουν διευρυμένοι ορίζοντες δηλαδή αναφερόμαστε πλέον και σε πρόσφυγες αλλά και σε ανθρώπους που προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδες κλπ. Ε, αυτό όμως θα γίνει του χρόνου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η συγκεκριμένη ε, πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τους πρόσφυγες. Αυτό θελήσαμε να προωθήσουμε και βάσει αυτό που μας ζήτησε και το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τώρα την κοινωνική ανάμειξη, δεν καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά την ερώτησή σας γιατί πρόκειται για projects τα οποία αφορούν ε, τους πρόσφυγες που θα παίξουν βεβαίως ε, με τα γειτονόπουλα, με τα παιδιά της γειτονιάς δηλαδή. Δεν ξέρω εάν ε, έχετε κάτι άλλο κατά νου. Σε αυτό το project πάντως δεν υπάρχουν ας πούμε ομάδες ποδοσφαιρικές που αποτελούνται αποκλειστικά από πρόσφυγες. Ε, ε, νομίζω ότι αυτό είναι το συγκλονιστικό ότι ε, μοιραζόμαστε στιγμές, μοιράζονται μάλλον στιγμές τα παιδιά είτε είναι πρόσφυγες είτε είναι τα παιδιά της γειτονιάς και ακριβώς επειδή μιλάμε σε συγκεκριμένα projects και για ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, ε, αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Ε, όσον αφορά την προώθηση της ε, ισότητας, ναι, είναι ένας από τους στόχους. Υπάρχουν projects για το κράινεμ, ναι, είναι το ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε και άλλα και άλλες ας πούμε αποκλειστικά γυναικείες ομάδες, πάλι με το ίδιο στυλ πρόσφυγες, μη πρόσφυγες. Ε, ε, ε, και ούτω ή άλλω δεν αναφερόμαστε μονάχα στο ποδόσφαιρο. Μιλάμε για τον αθλητισμό γενικότερα, έτσι ώστε να συμμετέχουν και γυναίκε και οπωσδήποτε αξιολογούμε στη διάρκεια τη αξιολόγηση του project και τα θέματα ισότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και έβαλα και τον εαυτό μου στην λίστα των αμιλητών. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσω με την συνάδελφο. Είδαμε διάφορα πλωτικά προγράμματα τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση και άλλοι συνάδελφοι θεωρούν ότι η ανταλλαγή στην διαδικασία αξιολόγησης με τους βουλευτές θα έπρεπε να είναι η επαφή με τους βουλευτές λοιπόν θα πρέπει να είναι πιο σωστή. Γιατί λείπουν κάποια στοιχεία. Για να μπορέσουμε σωστά να αξιολογήσουμε ένα έργο. Αυτό προφανώς και είναι φυσιολογικό γιατί κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα στο μέλλον να μπορέσουμε να έχουμε πιο στενή επαφή με τους ετούντες ε, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, να υπάρχει μια κάποια ανταλλαγή απόψεων, γιατί νομίζω ότι πολλά θέματα θα μπορούσαν να επιληθούν αν θα μπορούσαν να υπάρχουν ε, μία-δύο συνομιλίες σε αυτή τη φάση. Γιατί θα υπήρχε ανταλλαγή πληροφοριών. Γιατί στην τελική ανάλυση οι βουλευτέ καλούνται να τα καταλάβουν αυτά και να τα εξηγήσουν στου ψηφοφόρου του. Θα ήταν καλό λοιπόν να είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια τέτοια συνομιλία για να υπάρχει κάποια ανταλλαγή απόψεων μέσα στη φάση αξιολόγησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση και θα απαντήσω αυτά που είπα και προηγουμένως στην ε, συνάδελφό σας, την κυρία Κάμερ Εύερτ, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αντιτεθειμένη να έρθει σε επαφή με τους ετούντες και με τα σχετικά γραφεία κατά τη φάση της αξιολόγησης για να δούμε κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ε, για να δώσουμε συμβουλές σε ό,τι αφορά την κατηγοροποίηση στις εκάστοτε κατηγορίες Β, Α ή Γ. Τα τελευταία χρόνια κάναμε και κάποια ανημερωτικά σεμινάρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους βοηθούς, για τους ε, υπαλλήλου του Κοινοβουλίου για να εξηγήσουμε αυτό που σας εξηγήσαμε και εδώ σήμερα. Το ποια είναι τα κριτήρια, ποιες κατηγορίες υπάρχουν, τι θα πρέπει να προσέξει κανείς για να περάσει κάποιο πιλωτικό πρόγραμμα. Αν ε, εκφραστεί σχετικό ενδιαφέρον, μπορούμε να την ε, συνεχίσουμε αυτή την ε, παράδοση η οποία διακόπησε σε κάποιο σημείο και να κάνουμε λοιπόν ενημερωτικά σεμινάρια πριν από την προθεσμία υποβολή των αιτήσεων για το πώς κάνει την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποια είναι τα κριτήρια. Συγκεκριμένα τώρα, επειδή είπατε ότι οι συνάδελφοι στην Κομισιόν ενδεχομένως να μην γνωρίζουν, να μην έχουν ειδικέ γνώσεις για όλα τα θέματα, να σας πω ότι στην αξιολόγηση δεν εξετάζουμε την ουσία και την αξία των ε, προτινόμενων έργων, αλλά κάποια νομικά κριτήρια, κατά πόσον πληρούνται, για παράδειγμα, οι όροι του προγράμματος, της νομοθεσίας και του καθεξής. Ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα ότι ήμουν τελευταίος στον κατάλογο των ομιλητών, αλλά προσθέθησαν δύο συνάδελφοι. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είχα ζητήσει το λόγο, αλλά τέλο πάντων. Ε, έχω δύο ερωτήσεις. Ε, χαίρομαι για αυτό το μηχανισμό πιλωτικών σχεδίων. Εγώ είμαι νεοεκλεγμένη, είναι η πρώτη μου θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι σημαντικό να καταλάβω πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Έχω μια τεχνική ερώτηση. Ε, έχετε κάποια... Μπορείτε να δώσετε κάποια ενημέρωση για τους νεοεκλεχθέντες βουλευτές για να ξέρουν καλύτερα πώς πρέπει να κινηθούν και δεύτερον ποια είναι η προθεσμία για την επόμενη υποβολή προτάσεων. Ε, δεύτερον, ε, ερωτήσεις για συγκεκριμένα πιλωτικά σχέδια. Πρώτη ερώτηση αφορά το Music Moves in Europe. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό σχέδιο. Στην ε, παρουσίασή σας μιλήσατε και για εκπαιδευτικά θέματα. Αναρωτιέμαι, τα μουσικά σχολεία έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν σε αυτό το σχέδιο. Δεύτερη μου ερώτηση αφορά το την πρωτοβουλία για τον γραμματισμό για όλους. Είναι μεγάλη πρόκληση το να πλησιάσουμε τους ενήλικους που δεν βρίσκονται σε ένα, μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν υπάρχουν κάποια συμπεράσματα που βγήκαν από αυτό το σχέδιο, κάποιες καλές πρακτικές κλπ. Σας ευχαριστώ να δώσουμε το λόγο στους ε, προσκεκλημένους μας για να απαντήσουν. Για τα θέματα ενημέρωσης, ε, κάποιου σεμιναρίου ε, για τους νέους βουλευτές. Ε, αν το Ευρωκοινοβούλιο θέλει, πολύ ευχαρίστως. Τώρα σε ό,τι φορά το χρονοδιάγραμμα για, τα, για τις προτάσεις πιλωτικών προγραμμάτων, ε, ακολουθεί την διαδικασία του προπολογισμού, τη δημοσιοπική διαδικασία. Νομίζω ότι η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνει μέχρι το Μάιο και η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται τον Ιούνιο. Νομίζω ότι μπορείτε να ενημερωθείτε και από τη γραμματεία. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Media Literacy for All, για τους ενήλικους θα έλεγα ότι από την εμπειρία μας το πιο σημαντικό είναι να τους πλησιάσουμε μέσω υφιστάμενων φορέων μιας πόλης. Για παράδειγμα, μια συνεργασία ανάμεσα σε βιβλιοθήκες και οργανώσεις που ασχολούνται με το γραμματισμό, ε, όπου βιβλιοθήκες βοηθούσαν μεγαλύτερους ανθρώπους να γραμματιστούν με την χρήση προσωπικού εθελοντών νέων που βοηθούσαν τους γεραιότερους. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη δυνατότητα να πλησιάσουμε τους ενήλικους. Αλλά το καλό με αυτά τα σχέδια είναι ότι πάντοτε υπάρχουν και πρωτότυπες ιδέες, καινούργιες ιδέες που δεν είχαμε σκεφτεί στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ρικάρδο, θέλετε να πάρετε και εσείς το λόγο να απαντήσετε. Thank you very much for your question. Για το Music Moves Europe, να σας πω το εξή. Τα εκπαιδευτικά μαθήματα είναι ανοιχτά σε όλους. Και αυτούς φορείς που βρίσκονται και λειτουργούν μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και εκτός. Σας ευχαριστώ. Τελευταία ομιλήτρια. Φραγκόφσκι. Ε, Θα κάνω δύο ερωτήσει. Καταρχήν, σα ευχαριστώ πολύ για όλε τι λεπτομέρειε που μα δώσατε πολύ χρήσιμε πληροφορίε. Θα μπορούσατε να μα μιλήσετε λίγο περισσότερο για του υπότιτλου και το πρόγραμμα Arte στην τηλεόραση. Δεδομένου ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα τελειώσει του χρόνου με μεγάλη επιτυχία, υπάρχει πρόθεση να συνεχίσετε αυτή την πρωτοβουλία, να την επεκτείνετε στην ε, ε, επόμενη εκδοχή του προγράμματο Creative Europe. Και πώ θα μπορούσε να ενταχθεί μέσα σε, στην ε, νέα απόφαση που θα ληφθεί για τα προγράμματα. Ευχαριστώ. Thank you for your question. Πράγματι, είναι ένα εξαιρετικά πετυχημένο σχέδιο και όταν μια ομάδα παίζει καλά δεν την αλλάζεις. Ο προπολογισμός έχει αυξηθεί και έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσαμε να διευρύνουμε τα ωφελήματα που προκύπτουν από αυτό το σχέδιο. Θα πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν την ουσία του όπως έχει και να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να το περάσουμε σε άλλο επίπεδο. Δεν σκοπεύουμε όμως να... Δεν σκοπεύουμε, λέω, να αλλάξουμε την ουσία. Πρόκειται γιατί έχουμε ως πρόθεση να συνεχίσουμε στην ίδια άκουσα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ να κλείσουμε το θέμα λοιπόν αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, προσκεκλημένους μας. Βλέπετε πόσο μας απασχολεί το θέμα αυτό. Και ελπίζω μετά τη σημαντική ανταλλαγή αυτή που είχαμε να μπορέσουμε στο μέλλον να έχουμε πιο τακτικές ε, επαφές. Αυτό αποτελεί επιθυμία όλων των συναδέλφων. Θα θέλαμε λοιπόν να σας χαιρετήσουμε και προσβλέπουμε στην επόμενη ευκαιρία που θα έχουμε να συνομιλήσουμε μαζί σας. Liebe Kolleginnen und Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. Μία φορά το χρόνο τουλάχιστον στην Επιτροπή Πολιτισμού έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τους νέους Ευρωπαίους πολίτες. Και ο σκοπός μας λοιπόν είναι να λάβουμε υπόψη τις απόψεις, τις ιδέες, τις σκέψεις και τις ανησυχίες των νεαρών ανθρώπων για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συγκεκριμένες μας προτάσεις σε ό,τι αφορά και την διαδικασία λήψης αποφάσεων μας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική. Ένας βασικός μας πολιτι... ένα βασικό ε, εταίρος μας στην διαδικασία αυτή σε ό,τι αφορά την πολιτική για την νεολαία είναι το Ευρωπαϊκό Φόρουμ ε, Νεολαία. Ανδρέα Κασαμέτη και Γιούντι Λάντα εκπροσωπούν το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαία. Θα ήθελα να σα καλωσορίσω. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων λοιπόν έρχεται σε μια πολύ επίκαιρη χρονική στιγμή. Γιατί από ξέρετε έχουμε τα νέα προγράμματα για το Πουδουπού, τα οποία συζητιούνται ιδιαίτερα σε τρεμερεί διαλόγου με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα. Και όπω ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Σώμα αλληλεγγύης και το Erasmus Plus ε, προσανατολίζονται ιδιαίτερως στους νέους ε, πολίτες. Ε, πρόκειται για μια, νέα, για μια πρώτη ανταλλαγή απόψε με τα νέα μέλη λοιπόν της Επιτροπής μας και πριν από κάποιο καιρό είχαμε και τις ακροάσεις των νέων επιτρόπων. Πρόκειται λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ υλικό και ελπίζουμε ότι θα είναι πάρα πολύ συναρπαστική η συζήτησή μας. Χαίρομαι λοιπόν που θα ακούσουμε από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Επιτροπής ε, Πολιτισμού και ποιες πολιτικές προτεραιότητες ε, πιστεύετε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε για τους νέους ανθρώπους κατά την ε, θητεία αυτή. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για 15 λεπτά και μετά θα ακολουθήσει γύρω σε απαντήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που ξεκινάτε τον διάλογο αυτό μαζί μας και που βάζετε τους νέους στην επί... στο επίκεντρο της σημερινής σας συνεδρίασης. Έχουμε μακρά ιστορία εξαιρετική συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαία και χαιρόμαστε που είστε δεσμευμένοι για να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα για να βελτιώσουμε τη ζωή των νεαρών ανθρώπων, των ενανθρώπων. Πρωτού λοιπόν να ξεκινήσω, να σα αισθηθώ. Ανδρέα, ονομάζομαι και είμαι μέλο ε, του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Είμαι ένας από τους 11 θελοντές ε, που καθοδηγούν και διαχειρίζονται την οργάνωσή μας. Ε, έχουμε μαζί μας την Γιούντιτ Λαντάι και τον Αλφόνσο Γιούλιτ Λαντάι. Επίσης είναι ε, μέλη του προσωπικού μας. Ελπίζουμε να έχετε ερωτήσεις για να κάνουμε και μια συζήτηση μετά μαζί σας. Είναι η τιμή μα και χαρά μα που βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Πρωτού ξεκινήσουμε την ανταλλαγή απόψεων, να σας πούμε δύο λόγια για το ποιοι είμαστε. Εν συντομία, τι κάνουμε και ποιε είναι οι προκλήσεις των νέων ανθρώπων σήμερα. Και τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού για να δώσουμε απάντηση στις ανησυχίες αυτές. Να ξεκινήσω με την παρουσίασή μου λοιπόν για να δω λειτουργεί πολύ ωραία. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, μια ανεξάρτητη δημοκρατική οργάνωση η οποία καθοδηγείται από νέους ανθρώπους. Είμαστε, είμαστε μάλλον μια οργάνωση ομπρέλα. Έχουμε και μια γενική συνέλευση η οποία συναποτελείται από άτομα από τις ε, επιμέρους οργανώσεις μας. Εκπροσωπούμε τα Εθνικά Συμβούλια Νεόλεας. που είναι όλα μέλη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους νέους. Τι κάνουμε. Θέλουμε να δώσουμε πιο πολλές αρμοδιότητες στους νέους για να συμμετέχουν πιο πολύ στην ε, κοινωνική ζωή και να μπορέσουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους προς το συμφέρον ε, και των ε, νέων και των οργανώσεων. Ποια είναι λοιπόν τα μέλη μας, ποιες είναι οι οργανώσεις που είναι στην, στο φόρουμ μας. Έχουμε καταρχάς κάποιες οργανώσεις οι οποίες είναι και αυτές οργανώσεις που περιλαμβάνουν άλλες μικρότερες οργανώσεις. Μέσω του δικτύου λοιπόν αυτού έχουμε πρόσβαση σε εκατομμύρια νεαρούς ανθρώπους. Εκπροσωπούμε μια μεγάλη, ένα μεγάλο φάσμα νέων. ΛΟΑΔ, ΣΥΝ, νέοι στην Ήπεθρο, εθνικές μειονότητες και συνεργαζόμαστε επίσης και με άλλες οργανώσεις και πλατφόρμες που εκπροσωπούν που εκπροσωπούν για παράδειγμα νέους ε, Ρωμά, νέους μουσουλμάνους και άλλες ομάδες. Οι δράσει των μελών είναι επίσης πολύ ποικιλόμορφες ε, εργασία, εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτική εκπαίδευση, ε, αλλαγή του κλίματος, βιωσμή ανάπτυξη και ούτω καθεξή. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το φάσμα των δράσεων των μελών μας. Πρόκειται για μια οργάνωση που αυξάνεται αριθμητικά. Αυτό γιατί ο τομέας των νέων τονώνεται στην Ευρώπη. Οι νέοι όλο και πιο πολύ ενδιαφέρονται και θέλουν να συμμετέχουν ενεργά σε τέτοιε οργανώσει. Ένα σημαντικό παράδειγμα, βλέπετε ότι το Ευρωβατρόμετρο έκανε μία μελέτη τον Απρίλιο του φετινού έτου, η οποία καταδεικνύει ότι 75% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δραστηριοποιούνται σε κινήματα, σε δράσεις τέτοιες σε όλη τους ζωή. Και φυσικά τέτοιου είδους ε, συμμετοχή σημαίνει με τη σειρά τη ότι υπάρχει όλο και πιο μεγάλη υποστήριξη των δραστηριοτήτων των νέων. Χρηματοδότηση λοιπόν για τις οργανώσεις των νέων. Υπάρχει πιο πολύ χώρος ε, συμμετοχής ε, για τα νέα άτομα και μπορούν να συμμετέχουν πιο πολύ και να λαμβάνουν και στη διαδικασία έλλειψη αποφάσεων. Επίσης, οι νέοι, όλο και πιο πολλοί νέοι, ψηφίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πού φάνηκε αυτό? Στις ευρωεκλογέ που φανηκε αυτο στις ευρωεκλογες που εγιναν το 2019. Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ξεκάθαρα ότι η ηλικιακή ομάδα 18 μέχρι 24 ήταν αυκήνη που σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στα ποσοστά προσέλευσης στις κάλπες σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα 28% το 2014 σε 42% το 2019. Άρα προφανώς ήταν το κλειδί οι νέοι στις ευρωεκλογές του 2019. Παρ' όλα αυτά, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει υπερβολικά χαμηλή εκπροσώπηση των νέων στις διάφορες δομές για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Και εδώ είναι και ένα από τα βασικά μας ε, καθήκοντα. Προσπαθούμε να προωθήσουμε τη συμμετοχή των νέων στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η αύξηση της συμμετοχής των νέων στις ευρωεκλογές του 2019, εν μέρη οφείλονταν στο γεγονός ότι όλες οι οργανώσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιήθηκαν προς το σκοπό αυτό. Στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ, για παράδειγμα, νεολαία, κάναμε μια εκστρατεία, ενδεχομένω να την είδατε. Change is coming. Η αλλαγή έρχεται. Είχαμε ένα βαν, ένα φορτηγάκι το οποίο ταξίδεψε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σταματούσε σε πόλεις και κάναμε συνομιλίες με διάφορους νέους για την ευρωπαϊκή πολιτική και αυτό φυσικά ήταν μόνο ένα τμήμα της εκστρατείας μας και φυσικά δεν σταματήσαμε τη δουλειά αυτή μετά τις εκλογές, συνεχίσαμε. Συνεργαζόμαστε με πολλούς ευρωβουλευτές, για παράδειγμα, που έχουν μεγάλο πάθος για τη νεολαία δημιουργήσαμε μια νέα διακοινοβουλευτική ομάδα. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να χτίσουμε μια δυνατή τέτοια διακοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα θέματα που αφορούν του νέου εκπροσωπούνται σωστά σε όλε τι επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά λοιπόν εν συντομία σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαία. Να σα πω τι γίνεται τώρα με τι ανησυχίε και τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα. Γιατί μέσω των μελών μα μπορούμε να ρωτήσουμε του νέου τι είδου προβλήματα έχουν, τι είδου προκλήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα. Εδώ συμπεριλαμβάνουμε κάποιους από τους τομείς όπου οι νέοι θεωρούν ότι οι πολιτικοί ηθήνοντες θα πρέπει να αναλάβουν δράση. για να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα στη ζωή τους. Αλλά και του κλίματος και κρίση του κλίματος. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι θέλουν οι πολιτικοί να αναγνωρίσουν ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κρίσης και ότι θα πρέπει να αναλευθεί δράση βιώσιμη, μακροπρόθεσμη από τις, ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, από τις εθνικές κυβερνήσεις, προκειμένου να υπάρχει καν μέλλον για τους νέους. Βλέπουμε επίσης ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θεωρούνται πλέον ως κάτι πραγματικά δεδομένο τα δικαιώματα των νέων συχνά θεωρούν ε, οι νέοι ότι περιορίζονται, δεν υπάρχει σωστή πρόσβαση. Και μιλάμε για παράδειγμα για την πλήρη αξιοποίηση των δικαιωμάτων των νέων ε, από πολιτικά δικαιώματα, κοινωνικά, οικονομικά δικαιώματα. Επίσης, το γεγονός ότι συρρυκνούται ο, χώρο χώρος της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί πρόβλημα. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει συμμετοχή των νέων σε οργανώσεις, σε ακτιβιστικά κινήματα. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις. Υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα. Είναι πολύ περιοριστική σε κάποιες περιπτώσεις ε, η νόμοι που ενδεχομένως να τους ε, απαγορεύουν να συμμετέχουν σε κάποια κινήματα, σε κάποιες δραστηριότητε σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το σεξουαλικό προσανατολισμό τους, ΛΟΑΔΑ. Δημογραφικές ε, προκλήσεις προφανώς αποτελούν ένα ζήτημα γιατί ο πληθυσμός γυράσκει και Υπάρχουν πολλά εμπόδια, όπω σα είπαμε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των νέων στα δικαιώματά του, σε ό,τι αφορά την κοινωνική συμπερίληψη κτλ. Ξέρουμε ότι πολλοί νέοι θεωρούνται ότι είναι αποκλεισμένοι. Και τέλο, το θέμα τη ψηφιοποίηση. Εδώ η ψηφιοποίηση προφανώ επισέρχεται σε όλους τους τομεί τη σημερινή ζωή και αυτό έχει τι συνέπειε του. Τι κάνει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαία για να ανταποκριθεί στι προκλήσει αυτέ, πολλά. Πολλέ δράσει. Να αναφέρω κάποιε εξ αυτών. Έχουμε καταρχά το YoFest. Κάθε δύο χρόνια το διοργανώνουμε στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Εκδηλώσεων I 2018, για παράδειγμα. Βλέπετε ε, στο Στρασβούργο το YoFest ένα πολιτικό φεστιβάλ ε, το οποίο φέρνει σε επαφή τους νέους με τους πολιτικούς. 10.000 νέους ε, συγκεντρώσαμε στο Στρασβούργο την προηγούμενη φορά. Σκοπός μας είναι να κάνουμε μια συζήτηση για τις προκλήσεις και τη ζωή των νέων ανθρώπων. Επόμενη διοργάνωση 29 και 30 Μαΐου στο Στρασβούργο του χρόνου το 2020. Η Ευρωπαϊκή ε, Πρωτεύουσα Νεολαίες Κάποιες πόλεις ε, κάνουν αίτηση για να βελτιώσουν την πολιτική για τους νέους στην πόλη τους. Νόβησαν στη Σερβία, είναι η πόλη που επιλέχθηκε φέτος. Του χρόνου θα είναι μια πόλη στη Γαλλία. Και επίσης ένα άλλο πρόγραμμα είναι ο κατάλογος για την ε, πρόοδο της νεολαία, μια ανάλυση της ζωής των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, πέρα από τον οικονομικό, από την οικονομική διάσταση. Θα σας ε, πω και παραπάνω στοιχεία, αν θέλετε, για τα προγράμματα αυτά. Έχω τρία λεπτά ακόμα. Κάποια θέματα με τα, για τα οποία συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή Πολιτισμού. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εξαιρετική συνεργασία Erasmus Plus, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά με την κυρία Σέντροβα, την κυρία Φερέρα, με τους κοιοδοσίγητες και σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, ε, οι οποίες ανέφερα, ε, Γιώφεστ, Ευρωπαϊκός Πίνακας ε, Νεολαίας και εδώ θα χαρούμε ιδιαίτερως να συνεργαστούμε μαζί μας και να σας βοηθήσουμε με δικές μας δράσεις. Όπως σας είπα, τα προγράμματα αυτά είναι θεμελιώδη για τη ζωή των νέων και είναι σαφές ότι πρόκειται για προγράμματα που λειτουργούν ε, πολύ καλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρω... στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαία επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στα προγράμματα αυτά. Σε διάφορε περιστάσει αναφέραμε ποια είναι τα βασικά στοιχεία που μα αφορούν για το Ευρω... Erasmus Plus και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, να πω αν συντομία, θα θυμάστε ότι ζητάμε δεκαπλάσιο προπολογισμό και χαρήκαμε που το Κοινοβούλιο τριπλασίασε τον προπολογισμό. Είναι σημαντικό αυτό, προκειμένου να έχουν πιο πολλοί νέοι πρόσβαση στο πρόγραμμα αυτό και προκειμένου να υποστηριχθούν πιο πολλά προγράμματα νεολαία. Θέλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πραγματικά ανοιχτό σε όλους. Υποστηρίζουμε λοιπόν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καταστεί πιο συμπεριληπτικό το πρόγραμμα και επίση είναι σημαντικό επίσης να δούμε τι γίνεται και με την ε, κοινωνία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το Discover EU. Πολύ σημαντικό πρόγραμμα και αυτό που περιλαμβάνει και την διάσταση της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ε, εδώ λοιπόν υποστηρίζουμε τη διαδικασία εκμάθησης ε, των νέων και επίσης τι γίνεται με τη χρηματοδότηση του Discovery EU, μήπως είναι από άλλου τομεί που θέλουν και αυτή η χρηματοδότηση. Στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη χαιρόμαστε που υπάρχει επικέντρωση στην συμπερίληψη, στην προσβασιμότητα, μια ισορροπημένη πρόσβαση. Και επίση οι εθελοντικέ θέσει θα πρέπει να περιορίζονται σε μη κερδοσκοπικέ εταιρείε. Και τέλο, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την. Μάλλον εφαρμογή της στρατηγικής για τους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ για να υπάρχει σωστή αξιοποίηση των πόρων. Αυτά λοιπόν εισαγωγικά και τώρα με χαρά να κάνουμε μια συζήτηση, να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτό που με έκανε εντύπωση ε, στην παρουσίασή σας είναι πόσο σημαντικό είναι η νεολαία ναι, να έχει φωνή και να ακούγεται η φωνή της νεολαίας, της ευρωπαϊκής νεολαίας, να μπορεί να συμμετέχει. Και αυτό το λέω ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις, ε, την απόφαση για την μη έναρξη διαπραγματεύσεων με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Αυτό αποτελεί μεγάλη απογοήτευση για τη νεολαία. Ήμουν σε αποστολή παρατηρήσης των εκλογών στο Κωσυφοπέδιο και συνομίλησα με νέους οι οποίοι πραγματικά υπολογίζουν στην Ευρώπη, έχουν στραφεί όλος χερός προς την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το τελειφθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πόσο σημαντικό στοιχείο είναι η Ευρώπη για τους νέους. Και χαίρομαι λοιπόν όλος ιδιαίτερος που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Τσβέρ. Ευχαριστώ πολύ και για αυτή την συζήτηση. Είναι μεγάλοι φίλοι. η διαδικασία και πραγματικά θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία την οποία, της οποίας πρέπει να υπεραμεινθούμε και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο διάλογος με τους νέους πρέπει να είναι ευρύτερος όσον αφορά ε, το περιεχόμενο και θα πρέπει επομένως να ασχοληθούμε και ας πούμε και με τα θέματα ε, τα οικολογικά του κλίματος. Το ζητήσατε και εσείς άλλωστε. Βεβαίως καλύτερη χρηματοδότηση, ένας ευρύτερος προϋπολογισμός θα βοηθήσει στο μέλλον ε, την ε, οργάνωσή σας. Ξέρω ότι στην αρχή είσαστε πολύ αισιόδοξοι, είχατε πολύ αισιόδοξες έτσι, ε, αισιόδοξους προγραμματισμούς. Ε, επίσης ε, το Κοινοβούλιο επικρίθηκε γιατί προσπάθησε να τριπλασιάσει τον προϋπολογισμό. Αυτό όμως θα βοηθούσε την καλύτερη οργάνωση. Περισσότερα χρήματα, περισσότεροι πόροι σημαίνουν και μεγαλύτερη, μεγαλύτερες και περισσότερες σε ευκαιρίες ε, και για τους ε, νέους. Αυτό είναι ε, σαφές και θετικό αναφέρεται ότι θα πρέπει να παραμείνουν ε, οι παραδοσιακές δραστηριότητες ε, και πραγματικά ε, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές και να διατηρηθούν γιατί είναι πολύ σημαντικό και για το μέλλον. Εμείς θα εργαστούμε και με άλλες πανευρωπαϊκές οργανώσεις όπως υπόθηκε άλλωστε μαζικά συμμετείχαν οι νέοι στους ευρωπαϊκές εκλογές και αυτό έδωσε ένα καλό αποτέλεσμα όχι μόνο γενικά στην Ευρώπη, αλλά και ειδικά στη Σλοβενία. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε άλλε δύο ερωτήσει. Πέτρα. Ευχαριστώ πολύ. με Ανδρέα και αγαπητό Φόρουμ Νεολαία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας έχουμε μαζί μα σήμερα. Και να σα ευχαριστήσουμε όλο ιδιαίτερω για τι ε, ενέργειές σας, τις δράσεις σας τα τελευταία χρόνια και κυρίως για την καλή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Πολιτισμού. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και στο μέλλον. Πολλά σημαντικά θέματα αγγίξατε. Μία έκκληση έχω από πλευρά μου σε ό,τι αφορά το Erasmus Plus. Ζητήσαμε τριπλασιασμό των κονδυλίων. Είμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης και ακούμε κάποια πρωταριθμητικά στοιχεία από το Συμβούλιο και δεν προϊονίζουν ε, τίποτε καλό. Το Συμβούλιο ούτε διπλασιασμό δεν μας ε, δίνει των ε, ποσών και θα ήθελα να ακουστεί το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαία και στα άλλα κράτη-μέλη για να μα βοηθήσετε, να μα βοηθήσετε στον αγώνα μα αυτά για να πετύχουμε τριπλασιασμό των κονδυλίων. Γιατί νομίζω ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό και θετικό στοιχείο να το πετύχουμε, να μα καλύψετε τα νότα από πλευρά του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαία, να ξεκαθαρίσετε και στα κράτη-μέλη ότι η επένδυση στις νέου είναι επένδυση στο μέλλον και το Erasmus Plus χρειάζεται πιο πολλά χρήματα. Αυτό απευθύνω ως έκκληση για να μας καλύψετε. Ένα στοιχείο να αναφέρω. Μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα νεολαία η οποία είναι δυστυχώ λίγο στο, στη σκιά τη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού. Και είναι κρίμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικέ οι προτεραιότητε αυτέ που θέτετε και αυτά που προωθείτε. Πώ θα το προωθήσουμε αυτό το προϊόν, λοιπόν, αυτό, αυτή την ιδέα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και την εκτιμώ ιδιαίτερω. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Σόιτροβα. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση, αλλά κυρίως για τη συνεργασία. Όπως είπαν ο Μιλάν και η Πέτρα, θέλω και εγώ να θίξω το θέμα του προπολογισμού. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν ζητήσετε από τους ε, εταίρους σας από ε, του ανθρώπου με οποίου εργάζεται στα κράτη-μέλη να κάνουν τη δική τους καμπάνια, τη δική τους εκστρατεία ενώπιον των ε, εθνικών υπουργείων, των εθνικών υπηρεσιών για την αύξηση του προπολογισμού. Εδώ θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Αυτό θα ήταν μια κοινή δράση, ας πούμε, για τον προπολογισμό. Πρέπει να συνεργαστούμε πολύ στενά. Εσεί στο επίπεδό σα και εμεί στο δικό μα. Επίση, να θέσω το εξή ερώτημα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, που βρίσκεται, θέμα που βρίσκεται στον τριμερή διάλογο. Κατά τη διάρκεια του τριμερού διαλόγου, η Κομισιόν και το Συμβούλιο, τόσο εδώ όσο και στο Erasmus Plus, έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για την ε, κεντρική διαχείριση των ποσών. Ε, εμείς ε, θέλουμε οργανώσει όπως η δική σας να μπορούν να απευθυνθούν κατευθείαν και να υποβάλουν προτάσεις στην Κομισιόν και να μην μπαίνουν στο ίδιο καλάθι με μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. Η Κομισιόν δεν το δέχεται όμως. Δεν δέχεται να μπει κάτι τέτοιο στο νομοθετικό κείμενο. Για σας πόσο σημαντική είναι αυτή η πρόταση του Κοινοβουλίου. Ε, explain. Ευχαριστώ. Να σα δώσω το λόγο για να απαντήσετε τις ερωτήσεις. Καταρχήν ευχαριστώ για όλε αυτέ τι ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ για τι δικέ σα ευχαριστίες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή Κόλτ. Στο παρελθόν έχουμε πολύ ωφέλιμη και χρήσιμη, είχαμε πολύ ωφέλιμη και χρήσιμη συνεργασία και ελπίζουμε το ίδιο θα γίνει και κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία. Τώρα έχω Πολλέ σημειώσει μπροστά μου, αλλά θέλω να ξεκινήσω με το Erasmus Plus και τον προπολογισμό του. Άσφαλος, ο τριπλασιασμός του προπολογισμού είναι εξαιρετικά σημαντικός για το European Youth Forum. Στείλαμε πρόσφατα επιστολή προς όλους τους υπουργούς ε, των κρατών μελών και όχι μόνο των κρατών και όλων των χωρών που είναι μέλη μας. Τις επόμενες μέρες θα δείτε ότι θα δημιουργήσουμε και κάποια έτσι βαβούρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ε, για να εξαεξηγήσουμε τη σημασία του τριπλασιασμού. Όταν λέγαμε δέκα φορές Εράσμους, δεν ήταν ένα αστείο. Δεν το κάναμε για πλάκα, το κάναμε έτσι ώστε όλοι οι νέοι να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Και για να συμμετάσχουν όλοι οι νέοι χρειαζόμαστε δέκα φορές περισσότερα κονδύλια. Ο τριπλασιασμός βέβαια είναι ήδη σημαντικός και θα το στηρίξουμε. Ε, και σας βεβαιώ θα είμαστε πολύ παρόντες ε, και θα κάνουμε lobbying στις ενώπιον των κυβερνήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πάντοτε και είναι ακόμα ο πιο ισχυρό μας σύμμαχος σε αυτόν τον αγώνα για τον τριπλασιασμό των κονδυλίων. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα ε, Νέων, ο τίτλος δημιουργήθηκε πριν από 10 χρόνια. Και σε αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια είδαμε μεγάλες αλλαγές. Όλο και περισσότερες πόλεις ε, ζητούν τη διοργάνωση και μάλιστα και μετά το τέλος του χρόνου βλέπουμε ότι διατηρείται μεγαλύτερη χρηματοδότηση των οργανώσεων των νέων δίδεται μεγαλύτερος χώρος δράσης για αυτές τις οργανώσεις, οπότε δεν τελειώνουν όλα με το τέλος του έτους της Ευρωπαϊκής ε, Πόλης Νεότητας. Αυτός ο τίτλος ε, φέρνει άλλωστε και τους ε, θεσμούς, τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ πιο κοντά στους νέους και στους ανθρώπους, διότι αρχίζουν οι πολίτες και καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα πολύ Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι τα προγράμματα πώς εφαρμόζονται κλπ. Χαίρομαι που η Επιτροπή Καλτ ε, έχει αυτό το ενδιαφέρον θα μπορούσαμε να υποβάλουμε ένα πιλωτικό σχέδιο στο μέλλον, το λέω ως ιδέα. Πάντως, είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό τον τίτλο. Ε, για παράδειγμα, όταν μιλάμε για το Discover, Discover You ή για το Ευρωπαϊκό Σώμα Λεγγύης. Λέμε, εσείς που ταξιδεύετε, εσείς που προσπαθείτε να ανακαλύψετε την Ευρώπη, γιατί να μην σταματήσετε και στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων ε, ως μια στάση. Τι άλλο να πω τώρα... Κάτι για το Erasmus Plus και το Ευρωπαϊκό Σώμα αποκεντρωμένε Αποκεντρωμένες δράσεις. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ερώτηση. Είναι μία από τις πιο σημαντικές μας ανησυχίες, πιο σημαντικές διεκδικήσεις. Και πραγματικά, ειλικρινά μιλάω εκ μέρους των, όλων των μελών μας. Έχουμε πολλά ευρωπαϊκά δίκτυα, πολλές ευρωπαϊκές οργανώσεις που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα και προσφέρουν προσθέμενη αξία και πολύ συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση. Γιατί, για παράδειγμα, έχουν την έδρα τους στο Βέλγιο και ανταγωνίζονται με εθνικούς φορείς ε, για ποσά τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό αυτές οι οργανώσεις να μπορέουν να υποβάλουν τις προτάσεις κατευθείαν στην Κομισιόν. Όχι αποκεντρωμένα. Για παράδειγμα στο Erasmus Plus. Ευχαριστώ. So Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Άντερσον. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Έχω κάποιες ερωτήσεις να κάνω για να καταλάβω πιο καλά και την προσέγγισή σας. Καταρχάς, ε, γιατί πιστεύετε ότι οι νέοι δεν έχουν ε, ίση πρόσβαση στα δικαιώματά τους και δεν τους θεωρούμε πολίτες με, ίση, με ίσα δικαιώματα. Πού το στηρίζεται αυτό. Σε ό,τι αφορά ε, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει κάθε άτομο έναντι του κράτους. Τι εννοείται με την ε, παγκόσμια ηθαγένεια. Πώς ε, διαφέρει αυτό από την εθνική ηθαγένεια και πού είναι τα πλέον εκτίματα, σε τι μπορεί να ελπίζει βελτίωση ένα άτομο που έχει αυτή την διεθνή ηθαγένεια και σε ποιον, από ποιον πρέπει να ζητήσει τα δικαιώματά του αυτά. Ευχαριστώ. Κυρία Μελμπάρης, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι γιατί βλέπω και μια νέα γυναίκα από την Λετωνία εδώ, οπότε θα μιλήσω σε αυτή τη γλώσσα. Ε, σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις αυτές λοιπόν που ακούσαμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε εθνικό επίπεδο. Εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λοιπόν, ζητάμε πάντα να κοιτάξουμε τι μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Εσεί μα ζητάτε το αντίθετο. Τι μπορούμε να κάνουμε πιο πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο πολλά πράγματα από κοινού. Για μας λοιπόν είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε όχι μόνο για τους νέους, για τη νεολαία, αλλά και με τους νέους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για μεγάλο καθήκον, μεγάλη... μεγάλο τμήμα των καθηκόντων μας. Θα πρέπει να συναντιόμαστε λοιπόν με τους νέους. Και εγώ έχω κάνει ένα σχέδιο για το πόσα σχολεία μπορώ να επισκεφτώ στην Λετωνία. Τώρα, για το θέμα της παιδείας ε, σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό στην Λετωνία. Αυτό επηρεάζει προφανώς και τα κίνητρα που έχουν οι νέοι και τις δυνατότητες που έχουν να συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά έργα. Εδώ έχω να σας κάνω μία ερώτηση. Τι περιμένετε από εμά, τι θέλετε να κάνουμε σε εθνικό επίπεδο, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε εθνικό επίπεδο. Η κυρία Πεντζαμία έχει το λόγο. Gracias, Ευχαριστώ. Καλώ ήρθατε στην Επιτροπή Κούλτ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σα. Τρία πράγματα. Μια ερώτηση για το πώ χρηματοδοτήσετε εσεί οι ίδιοι και τι προπολογισμό έχετε. Δεύτερον, αναφέρατε διάφορε προκλήσει για τους νέου στην Ευρώπη. Εγώ Μιλώ πιο πολύ βλέποντας τα πράγματα από την Ισπανία, αλλά δεν γίνεται πολλής λόγος για την απασχόληση των νέων και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι να βρουν μια θέση εργασία, καθώς επίσης και την ε, πρόσβαση στην στέγη. Επίσης δεν κάνατε λόγο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν προκειμένου να γίνουν επιχειρηματίες, να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώ δεν πρόκειται για προτεραιότητε για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο είναι μόνο για την Ισπανία. Γι' αυτό δεν ξέρω. Εσεί θα μου πείτε. Επίση, ε, λέμε, λέτε συνεχώ πρέπει να διευρυνθεί ο προπολογισμό, να αυξηθεί ο προπολογισμό για όλε τι πρωτοβουλίε. Συμφωνώ, είναι σημαντικέ οι πρωτοβουλίε αυτέ. Θα ήθελα να σα ρωτήσω όμω, ποιος είναι ο δικός σας ρόλος για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση για να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας ε, στην Ευρώπη για να διευρυνθεί το κράτος πρόνοιας, για να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες. Ε, ποιος είναι ο δικός σας ρόλος σε όλη αυτή τη διαδικασία του ευρωπαϊκού οράματος. Ευχαριστώ. Äh, να ακούσουμε, αφού ακούσαμε τρεις ερωτήσεις, να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Yes, thank you very much once again. Uh, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ε, βγαίνουμε λίγο από το, την, ε, τη ζώνη στην οποία αισθάνομαι πολύ άνετα να απαντήσω. Πάνω θα προσπαθήσω. Ε, σας με ρωτήσετε τι κάνουμε σε εθνικό επίπεδο. Ε, πηγαίνετε στη Λετωνία, στο Συμβούλιο των Νέων της Λετωνίας, στις εθνικές οργανώσεις, μιλήστε με τους ε, νέους, ε, δώστε τους το λόγο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Επίσης η συμβουλή μου είναι ότι ακούτε φέρνετε τα πίσω εδώ. προκειμένου να ληφθούν υπόψη. σε ό,τι αφορά το πόσο ίσοι μεταξύ τους είναι οι νέοι ως πολίτες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα προφανώς είναι καθολικά. Εμείς αυτό που διεκδικούμε είναι όλοι οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Για παράδειγμα, πρόσβαση σε θέσεις, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης ή σε στέγαση. Θα μπορούσαμε να τα αναφέρουμε ένα προς ένα, αλλά δεν έχει νόημα. Το θέμα λοιπόν θα έπρεπε να είναι αυτό. Η δυνατότητα οι νέοι να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους ε, Γιατί βλέπουμε πολύ συχνά αρνητικές διακρίσεις εναντίον των νέων εξαιτία ηλικία τους καθώς επίσης ε, και δυσκολίες πρόσβασης ε, στις ε, κοινωνικές πολιτικές και στο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Για παράδειγμα, κάποιοι νέοι δεν έχουν δικαίωμα να είναι δικαιούχοι συγκεκριμένων ενισχύσεων, κονδυλίων ε, κλπ. εξαιτίας ηλικία τους. Οπότε τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά και γι' αυτό μιλάμε. για την άσκησή τους ε, γενικά. τώρα να επιταχύνω λίγο. Το θέμα της ε, απασχόλησης είναι πολύ σημαντικό. Και στη δική μου χώρα, την Ιταλία, όχι μόνο στην Ισπανία. Άλλωστε το βλέπουμε και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το είπα εντάχει αλλά είναι πραγματικά προτεραιότητά μας. Για παράδειγμα, έχουμε συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα της εγγύησης για τους νέους, το Youth Guarantee. Επίσης, για το θέμα ε, των περιόδων μαθητείας, άμυστων περιόδων ε, μαθητείας, ε, για το οποίο συνεργαστήκαμε με την διακομματική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου. Ε, υπάρχει ένα θέμα στο Βέλγιο. Θέλουμε να απαγορευτεί σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου και του Βελγίου, αυτή η πρακτική των άμυστων ε, περιόδων μαθητεία. Εργαζόμαστε λοιπόν σε διάφορα θέματα και με διάφορους τρόπους για να καλύψουμε και αυτό το ζήτημα. Τώρα, το πώς χρηματοδοτούμαστε. Δυστυχώς, ομολόγω δεν έχω ακριβώς το νούμερο. Α, όχι, μου το, δείχνει, μου το δίνει η Λίμπα. Χρηματοδοτούμαστε κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή βασικά. Ο προπολογισμό μας είναι περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ το έτος. Έχουμε κάποια χρηματοδότηση και από το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, και ε, έχουμε και έσοδα από τα ίδια μας ε, τα μέλη, τα οποία πληρώνουν συνδρομές. Ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας έχει χρηματοδοτήσει για το UFEST, το φεστιβάλ το οποίο σας έλεγα προηγουμένως. Οπότε έχουμε ε, χρηματοδότηση από διάφορες πηγές, όμως το μεγαλύτερο τμήμα προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε κατά βάση μια ανεξάρτητη πλατφόρμα και προσπαθούμε να γίνουμε όσο, πιο, όσο πιο βιώσιμοι γίνεται με τον χρόνο. Νίκλας, ich gebe dir das Wort. Νίκλας, να πάρεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Και που προωθείτε αυτή την ε, διακοινοβουλευτική ομάδα για την νεολαία και ήμουν από αυτούς που υποστήριξαν ε, την ομάδα και πιστεύω ότι και η συμμετοχή θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Έχω κάποιες ερωτήσεις να κάνω για την Ευρωπαϊκό Πίνακα Νεολαίας. Σε ό,τι αφορά επίσης την ιδέα για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα αν θέλουμε να βγει από το πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού, να ε, κάνουμε αυτό που κάνουμε και στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμική Πρωτεύουσα, να επισκεφτούμε από πλευρά της Επιτροπής Πολιτισμού της ε, Πρωτεύουσας Νεολαίας. Να πω επίσης το εξή. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς θα προωθήσουμε τις δράσεις μας. Για παράδειγμα, έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Νεολαία. Αυτό είναι λίγο πιο πολύ ένα σοου, δεν έχει τόσο πολύ ουσία. Θα μπορούσαμε να θεσμοποιήσουμε την συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάποιας μορφής, κάποιου είδους κοινοβουλευτικών ομάδων ένα κοινοβούλιο για την νεολαία, για παράδειγμα. το οποίο θα εισακούεται και θα μετράει η φωνή του. Να μην είναι μόνο για το σοου ή το Θεαθήνα. Danke. Herr Sie haben Ο κύριος αλλά παρακαλώ να μην ε, υπερβείτε το χρονικό όριο. yes. Uh, <clears throat> very Ευχαριστώ πολύ κύριε Κασαμέντη για την παρουσίασή σας. Για τα πολύ σημαντικά στοιχεία που μας δώσατε, που λέτε ότι η συμμετοχή των νέων έχει αυξηθεί κατά 14%, από το 28% στο 42%. Μπορείτε να μας πείτε αν αυτή η αύξηση ε, έχει προκύψει πιο πολύ για τα φιλοευρωπαϊκά ή για τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα. Επίσης για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Γνωρίζετε ότι το διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Επί τη ευκαιρία συμφωνώ με τη Μαρία Σεντρόβα και με την κυρία Καμενεβέρτ για όσα είπανε. Πιστεύετε όμως ότι χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση το πρόγραμμα αυτό. Με, και με ποια δικαιολογία, με ποια αιτιολόγηση. Η euh, κυρία Γενμπού, Όπως γνωρίζετε, διαπραγματευόμαστε το νέο πρόγραμμα Εράσμους και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οι στόχοι της, ε, των προγραμμάτων αυτών θα πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνουν ε, τον εθελοντισμό, την εργασία με τους νέους, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα ένταξης μεγαλύτερων ομάδων του πληθυσμού οι οργανώσεις νέων θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ε, να πλησιάσουν αυτές τις ομάδες στόχους. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε λίγο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ως οργανώσεις στην ένταξη, στην ενσωμάτωση. Πώς μπορούν αυτά τα προγράμματα να φτάσουν στους ε, πιο αποκλεισμένους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σα. Όλο όσο πιο πολύ γερνάει κανένα, τόσο λιγότερο καταλαβαίνει του νέου. Οπότε <laughs> πολύ καλά που είσαστε εδώ μαζί μα. Ε, έχω τι εξή πρακτικέ ερωτήσει. Πρώτον, επισκέφθηκα την ιστοσελίδα σα. Δεν βλέπω όμω εκεί ένα κατάλογο με όλες τις ενώσεις, τα μέλη σας, γιατί λέτε ότι έχετε ένα πολύ μεγάλο αριθμό οργανώσεων στην πλατφόρμα σας. Θα ήθελα να μπορέσω να έρθω σε επαφή με κάποιες από αυτές. Δεύτερον, διευκρινήσεις για το πώς πλησιάζετε τους νέους. Ε, οι νέοι ε, μας εξέπληξαν με την κινητοποίησή τους για τις ευρωπαϊκές εκλογές, για την κλιματική αλλαγή κλπ. Αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι μαγειρεύεται εκτός του θεσμικού ραντάρ. Εσείς είστε εδώ σήμερα, αλλά πολλά πράγματα γίνονται ε, εκτός ευρωπαϊκών θεσμών. Έχετε κάποια στοιχεία να μας δώσετε για το τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ. Και τώρα να ακούσουμε τι απαντήσεις. Yes, thank you very much. Mm, so, the... ο, ο δείκτης ε, ε, πρόοδου της νεολαίας. Το σημαντικό με αυτό το δίκτυο είναι ότι μετρά την ποιότητα ζωής των νέων. Εξετάζουμε τρεις βασικούς δείκτες. Οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες, ε, οι ευκαιρίες και η βάση της ευημερίας. Δηλαδή δεν μετράμε οικονομικά στοιχεία, οικονομικούς δείκτες, δεχόμαστε ως βάση αυτά τα τρία στοιχεία, αυτές, αυτές τις ε, τρεις ιδέες. Πιο συγκεκριμένα έχουμε 60 υποδείκτες. Ένα από τα βασικά πορίσματα είναι ότι όσο περισσότερος χώρος υπάρχει για τις οργανώσεις νέων σε μια χώρα, τόσο πιο μεγάλη είναι η τόσο πιο ψηλό είναι ο δείκτης πρόοδου. Και αυτό ίσως θα μπορούσαμε να σας το εξηγήσουμε με περισσότερε λεπτομέρειε κάποια στιγμή, αλλά μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα μας. Εύκολα βλέπετε όλα τα συμπεράσματα τα οποία βγάλαμε μέσω της ε, υιοθέτηση του δείκτη αυτού που δεν κοιτάει οικονομικά δεδομένα, ΑΕΠ κλπ. Η συσχέτιση του δείκτη με το ΑΕΠ όμως δείχνει ότι χώρες με παρόμοια επίπεδα ΑΕΠ μπορούν να έχουν πολύ διαφορετικούς δείκτες, δηλαδή πολύ διαφορετικές τιμές του δείκτη. Έχουμε σημαντικά συμπεράσματα που βγήκαν και Πιστεύω ότι θα μπορούσατε να είναι και για σας πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά να τα χρησιμοποιήσετε. Σε ό,τι αφορά την συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ομάδων νέων. Η δική μας αποστολή είναι προφανώς να είμαστε η φωνή των νέων στην Ευρώπη και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε μαζί σας πολύ πρόθυμα. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός που είναι η συνδιαχείριση. Ακούγεται παράξενα, αλλά στην πραγματικότητα στόχος είναι οι νέοι να έχουν τις ίδιες δυνατότητες λήψης απόφασης με τις κυβερνήσεις, με τους αρμόδιους επίσημους φορείς στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Πάντως χρειαζόμαστε πιο τακτική και πιο διαρθρωμένη συμμετοχή. Το να οργανώνουμε κατά καιρού εκδηλώσεις είναι καλό, αλλά χρειάζεται κάτι πιο διαρθρωμένο, όπως έναν διαρθρωμένο διάλογο με φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω ακριβείς πληροφορίες για το πώς ψήφισαν οι νέοι, αλλά μπορώ να βρω αυτά τα στοιχεία και να σας τα στείλω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Ελληνικής, σίγουρα πιστεύουμε πως χρειάζεται κατάλληλη χρηματοδότηση προκειμένου να εξασφαλίσουμε ποιοτική δράση. Αν δούμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ορανώσεις που εργάζονται ποιοτικά και δεν έχουν ως στόχο απλώς να αυξήσουν τον αριθμό των νέων που πηγαίνουν από μια χώρα στην άλλη, τότε πρέπει να τις χρηματοδοτήσουμε. Το να επενδύσουμε στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι σαν να επενδύουμε στην κοινωνία των πολιτών και σίγουρα δεν μπορεί να είναι λάθος, δεν μπορεί να είναι σφαλμένο. Μετά, για τις μειονεκτικές ομάδες, μειονεκτούσες ομάδες και το Erasmus+. Plus. Είναι βασική μας διεκδίκηση. Εδώ και χρόνια. Από όταν ξεκινήσαμε τη δουλειά μας για το Erasmus+. Plus. Ζητούμε κατάλληλη χρηματοδότηση για να ξεπεράσουμε όλων των ειδών τους φραγμούς. Ένας νέος μπορεί να αντιμετωπίσει πολλούς διαφορετικούς φραγμούς και να, που δεν του επιτρέπουν να συμμετάσχει σε μια διαδικασία κινητικότητας. Μπορεί να είναι φραγμοί που έχουν σχέση με την κατάσταση, σωματική του κατάσταση, μπορεί να έχουν σχέση με τις γλωσσικές του ικανότητες κλπ. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήλθατε, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σα για την παρουσίαση που κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να επεκτείνουμε τη συμμετοχή των νέων, να την ενισχύσουμε. Είναι σημαντικό για όλη μας την κοινωνία και για το μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ. Ελπίζω να σας δούμε σύντομα και να είμαστε σε τερική επαφή. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nun geht es mit dem nächsten Punkt weiter. ευχαριστώ να περάσουμε στο επόμενο σημείο στη μερική διάταξη, λέει ο Πρόεδρος, σε ό,τι αφορά την παρουσίαση των ε, νικητών του Ευρωπαϊκού α, Βραβείου για την Εωλία. Είναι παράδοση πλέον η Επιτροπή Πολιτισμού να καλεί τις τρεις ομάδες νικητών του, του Ευρωπαϊκού βραβείου αυτού για την νεολαία για να μας παρουσιάσουν τα έργα του και χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που έχουμε μαζί μας τις τρεις ομάδες των ε, νικητών το 2019 από την Ιταλία, Φιλανδία και Αυστρία. Σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Ελπίζουμε να έχουν καταστάσει. you. Ich stelle jetzt ganz kurz... Äh, Να κάνω μια σύντομη παρουσίαση των ε, νικητών. Να ξεκινήσουμε με τον Φαμπιάνο Κατάνια και την Αλύση Πλάτα από την Ιταλία που θα παρουσιάσουν το έργο Eurofonica, το οποίο τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο μετά την Ιντα Αερόλα και τη Βίλα Γιάρα με το έργο European Citizenship του Ευρωπαϊκού α, Κοινοβουλίου των Νέων της Φιλανδίας. Δεύτερο βραβείο έλαβαν. Και στη συνέχεια έκαναν Γιάσαρ και η κυρία Ζένε Μπούχρα από την Αυστρία, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το έργο «Μουσουλμάνοι κατά του αντισημιτισμού» που βραβεύτηκε με το τρίτο βραβείο. Οι δύο αυτές νέες ε, κάθονται στο Προεδρείο, δεν χωράνε όλοι, γι' αυτό λοιπόν θα τους διαδοχικά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τρίτο βραβείο. Η κυρία Γιάζαρ και η κυρία Πούχρα από την Αυστρία. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεολαία που μας ε, επιτρέπει να παρουσιάσουμε σήμερα το βραβευμένο μας έργο «Μουσουλμάνοι κατά του αντισημιτισμού» που θέλουμε να ευαισθητοποιήσει τους μουσουλμάνους για να κατανοήσουμε τον αντισημιτισμό, αλλά όχι μόνο τον κατανοήσουμε, αλλά και να τον καταπολεμήσουμε. Έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό εδώ και χρόνια. να δούμε τις διαφάνειες. Σκοπός μας είναι λοιπόν να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους ε, μουσουλμάνους και έχουμε χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους προς την κατεύθυνση αυτή για την καταπολέμηση ε, του φαινομένου του δεσμετισμού και την κατανόηση του από διάφορες οπτικές, οπτικές γωνίες. Ευαισθητοποίηση λοιπόν ε, επικεντρωνόμενη στην κατάρτιση. Τρεις βασικούς πυλώνες έχουμε. Κατάρτιση, συναντήσεις και ανάμνηση. Γιατί αυτό μας επιτρέπει βιώσιμα να επιστητοποιήσουμε και να επηρεάσουμε τους νέους κατά του αντισημιτισμού. Χρειάζεται λοιπόν κατανόηση, αλλά χρειάζεται και επαφή και γνωριμία με την εβραϊκή κοινότητα. Για να γνωρίζουμε ποια είναι η ιστορική ευθύνη των νέων Ευρωπαίων το κομμάτι της κατάρτισης το έχουμε αναπτύξει με διάφορες ε, εκδηλώσεις, σεμινάρια, ε, workshop ε, διαφόρων εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με τον αντισημιτισμό. Το συνδέουμε και με τις ιστορικές ρίζες του ασημιτισμού, αλλά και με την σημερινή μορφή του αντισημιτισμού. Και βασικά ένα βασικό στοιχείο του έργου εστιάσατε και στη δημιουργία ευκαιριών συνάντησης μεταξύ μουσουλμανικής και ιουδαϊκής κοινότητας. Προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση και από τις δύο πλευρές. Έχουμε καλέσει λοιπόν εξέχουσες ε, εβραϊκές ε, προσωπικότητες οι οποίοι και ήρθαν στις εκδηλώσεις αυτές για να υπάρχει συνάντηση όχι μόνο με εβραϊκά, εβραϊκές προσωπικότητες, αλλά και με συναγωγές, με μουσεία. Όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά. Και η μνήμη δεν έχει να κάνει μόνο με την ίδια την ιστορία προφανώς, αλλά και με τη δημιουργία σύνδεσης με τη σημερινή κατάσταση. Δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε να μην ε, συμβεί ποτέ ξανά κάτι τέτοιο. Ανταστρέψουμε το βλέμμα μας στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον. Και αυτό θεωρώ ότι αποτελεί και βασικό τμήμα της εκπαίδευσης σχετικά με το ολοκαύτωμα. Είχαμε την μεγάλη τιμή να συνομιλήσουμε με επιζώντα ε, της, ε, του στρατοπέδου συγκέντρωσης και ήταν η πρώτη φορά που ήλθε η συγκεκριμένη κυρία σε μουσουλμανική κοινότητα. Διοργανώσαμε μια εκδήλωση, μια επίσκεψη πολυμερή πολλών ημερών για την ε, επίσκεψη στα μέρη αυτά και συνεργαστήκαμε με διάφορες άλλες υπηρεσίες και το έργο έκλουσε με μια μεγάλη καταληκτική εκδήλωση με πολλά μέλη της Ιουδαϊκής κοινότητας. Συμμετείχαν επίσης πολλά μέλη της ε, μουσουλμανικής κοινότητας. Δεν υπήρχαν στο παρελθόν τέτοιε εκδηλώσει. Γι' αυτό χαρήκαμε που υπήρχε θετική αξιολόγηση. Δυστυχώ. Βραβευτήκαμε με το βραβείο Κάρλ, λοιπόν, ε, Κάρλος. Ο Λουίτζι Τοσκάνο, ο φωτογράφος, ε, διοργάνωσε μία έκθεση στη Βιέννη και παρουσίαζε πορτρέτα α, επιζώντων και τρεις φορές έγιναν επιθέσεις κατά της εκδήλωσης αυτής. Μόνο στη Βιέννη υπήρξαν τέτοιε επιθέσεις. Κινητοποιηθήκαμε λοιπόν και είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν και στη χώρα μας δεν χωράει αντισημιτισμός και ρατσισμός. Κάναμε λοιπόν μια... Πήραμε μια απόφαση με άλλες ε, οργανώσεις και αποφασίσαμε νύχτη μερών να φυλάμε την έκθεση αυτή. Ήρθαν και άτομα από εβραϊκές ε, οργανώσεις, ε, ραβίνοι, μας έφεραν φαγητό ζεστά Δημιουργήθηκε λοιπόν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα παρά την ε, πολύ επιθετική πρόκληση τέτοιων φαινομένων και νομίζω ότι μαζί καταφέραμε να δείξουμε ότι δεν επιτρέπονται τέτοια φαινόμενα στην όμορφη Αυστρία μας. Ήταν λοιπόν εξαιρετική αυτή η εμπειρία και μας έδειξε πώς μπορούμε να ε, δώσουμε το στίγμα μας με τέτοιες εκδηλώσεις και στο μέλλον. Αυτό λοιπόν ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την κατανόηση από πλευρά μα και νομίζω ότι ήταν και ένα σημαντικό, μια σημαντική ένδειξη και για την εβραϊκή κοινότητα στην Αυστρία αλλά και σε όλον τον κόσμο. Ήταν άτομα που ήρθαν και μα είπαν: Κοιτάξτε, ήρθαμε το αεροπλάνο, γιατί τόσο σημαντικό ήταν το θέμα αυτό για μα. Και όλα αυτά δημοσιεύτηκαν και σε ένα μεγάλο άρθρο. Και δεν θα πρέπει να υποτιμάμε λοιπόν πόσο σημαντική είναι και η συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα Η Καταρίνα Φων Σνούρ δραστηριοποιείται για τον αντισημετρισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατάλαβε γρήγορα τι σημασία έχει αυτό το έργο για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ήρθε και στη Βιέννη μάλιστα αεροπορικός να μας επισκεφτεί και πραγματικά αναγνώρισε κατευθείαν την αξία του έργου μας και μας κάλεσε σε διάφορες περιστάσεις ε, για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα αυτό ως ένα παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ευρώπη. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και πολλοί άλλοι πρέσβεις μας υποστηρίξαν πάρα πολύ από την πρεσβεία της Αμερικής. Αυτά λοιπόν ήθελα να αναφέρω για τη βιωσιμότητα τώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το έργο μας. Θέλουμε να ξεκινάμε έργα βιώσιμα, τα οποία θα έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Και γι' αυτό χάρηκα που έχουμε και μία δημοσίευση, ένα εγχειρίδιο δημοσιεύτηκε για το έργο μας, όπου συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλά άρθρα των εμπειρογνωμόνων που συνεργάστηκαν, που έκαναν, συνέβαλαν. Και αυτό θεωρώ ότι θα αποτελέσει και ένα πρότυπο για διάφορες άλλες οργανώσεις, για την διοργάνωση τέτοιων έργων, προκειμένου να υπάρχει πραγματικά στοχευμένη αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και για τις ΜΚΟ θα μπορούσε να χρησιμεύσει αυτό το εγχειρίδιο. Σήμερα έχω μαζί μας, έχουμε μαζί μας και διάφορα τέτοια εγχειρίδια. Αν θέλετε, με χαρά να σας τα δώσουμε. Δυστυχώς ε, είναι στα γερμανικά, αλλά έχουμε και ένα φυλάδιο στα αγγλικά. Αυτή είναι επίσης η εταίρη μα με τους οποίους και συνεργαστήκαμε. Έχουμε πολλούς εβραϊκούς ε, τέτοιους ε, οργανισμούς, αλλά και πρεσβείες, όπως σας είπαμε, και το καθεξής. Αυτά από πλευράς μας. Και με χαρά θα ακούσω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Meine Hochachtung und mein Respekt. Σας εκφράζω το θαυμασμό μου και το σεβασμό μου για την ε, συμβολή του έργου σας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και ξέρω γιατί μιλάω. Η μητέρα μου επέζησε του ολοκαυτώματος και το γεγονό ότι τώρα ξεκινάει αυτό το έργο καταδεικνύει πόσο επίκαιρα είναι ακόμα τέτοια ζητήματα. Και γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητα τέτοια έργα, τέτοια προγράμματα όπως το δικό σας για μια κοινωνία η οποία θα αποτέχεται τη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία. Να δώσω τώρα την ευκαιρία στους συναδέλφους να κάνουν ερωτήσεις. Να είστε παρακαλώ συνοπτικοί, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Η Πέτρα. Δεν θέλω να κάνω οποιαδήποτε ερώτηση. Να πω ένα ευχαριστώ, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικό το πρόγραμμα και δυστυχώς εξακολουθεί να είναι απαραίτητο. Είναι πάρα πολύ όμορφο, θεωρώ, το γεγονός ότι οι γυναίκες μουσουλμάνες αναλαμβάνουν αυτό το καθήκον, το οποίο δεν ήθιστε. Ίσως να είναι και πρωτάκουστο σε αυτή τη μορφή. Συχνά είναι Αυστριακοί, Γερμανοί οι δράστες αυτοί που αναλαμβάνουν τέτοιες ε, ε πρωτοβουλίες. Αλλά τώρα είναι μουσουλμάνοι, μουσουλμάνες αυτές ε, οι γυναίκες που ξεκινούν τη διαδικασία αυτή και την πρωτοβουλία αυτή. Για να μην υπάρξει αντισημιτισμός. Γιατί ο αντισημιτισμός δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Πολύ απλό. Όπως ε, επίσης δεν ε, δικαιολογείται να έχουν θέσει οποιαδήποτε αντιμουσουλμανικά συναισθήματα ε, και εκδηλώσει στην κοινωνία μα. Γι' αυτό λοιπόν σα ευχαριστώ όλου ιδιαίτερω από το βάθο τη καρδιά μου και ελπίζω να συνεχίσετε το έργο σα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βραβείο Νεολαία ήταν μεγάλη αναγνώριση για μα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σα. Είναι σημαντικό επίση θεωρώ να κάνει ο καθένα αυτό που του αναλογεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για μα αυτό αποτελεί κάτι αυτονόητο. Και θεωρούμε ότι έχουμε την ευθύνη μας όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Η κυρία Σόντροβα. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου. Κυρίως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σας διότι ξεκινήσατε αυτό το ε, project ε, χωρίς να ξέρετε φυσικά ότι ε, θα λαμβάνατε αυτό το βραβείο. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να καταπολεμηθεί ο αντισημιτισμός. Είναι απαραίτητο να υπάρχει και διαθρεσκευτικός διάλογος. Γι' αυτό εκτιμώ ιδιαίτερος την πρωτοβουλία σας και ελπίζω ότι θα ε, εξεκολουθήσει αυτή η προσπάθειά σας να στέφεται από επιτυχία και να έχει νόημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γελμα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ ε, εκτός από τα συγχαρητήρια να εκφράσω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και ευελπιστώ ότι θα αποτελέσει ένα απλό ξεκίνημα, ένα έναυσμα. Ε, λυπούμε όμως γιατί δεν μπορώ να διαβάσω το βιβλίο σας, ε, είναι γραμμένο στα γερμανικά, δεν διαβάζω δυστυχώς την γλώσσα αυτή και ρωτώ πώς είναι, θα ήταν δυνατόν να μεταφραστεί το βιβλίο αυτό και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Θα μπορούμε μπορούσαμε να συμβάλλουμε, υπάρχει κάποιο είδος συμβουλής, διορθώνω, συμβολής ε, ε, στο μεταφραστικό έργο ε, και απευθύνω την ερώτηση και σε όλους τους υπόλοιπους παρισταμένους βουλευτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο προβουλευτές. Συγγνώμη να βγάλω τα ακουστικά μου λίγο, την μπερδεύομαι. Η ιδέα της μετάφρασης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή. Ίσως θα μπορούσαμε να λάβουμε ε, κάποια χρηματοδότηση, γιατί αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πιστεύω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τους επένους σας. Ε, θεωρώ ότι το project μόλις έχει ξεκινήσει έξι μήνες μόνο και δεν ξέραμε πώς θα την δράσει ο κόσμος. Είναι πραγματικά ένα θέμα σοβαρό. Αλλά ήταν σημαντικό, το προωθήσαμε με θάρρος και περιμένουμε να δούμε τι θα μας φέρει το μέλλον. Αν Και εγώ θα ε, σας ευχαριστήσω για την προσπάθειά σας. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πρόσφατα αναφερθήκαμε στην ε, απόπειρα που έγινε κατά του τζαμιού στο Χάλ Είχαμε και πρόσφατα τις προηγούμενες μέρες μια ε, αντίστοιχη επίθεση. Σας ε, ευχαριστώ και σας συγχαίρω ε, για αυτήν την προσπάθειά σας. Εγώ προσυπογράφω και την ιδέα της μετάφρασης του βιβλίου. αλλά και μια ερώτηση, μια και είμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε σχέσεις με άλλες οργανώσεις μουσουλμανικές έτσι ώστε ε, να συνεχίσετε και να διευρύνετε το σχέδιο που έχετε ξεκινήσει. Στην παρούσα φάση δεν έχουμε ακόμα επαφές με άλλες διεθνείς οργανώσεις νέων. Αλλά θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν ξέρω κατά πόσον θα είχε νόημα να ανταλλάξουμε στοιχεία για να έχουμε ένα δίκτυο σιγά σιγά επαφών. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστούμε την κυρία Γιάννη, την κυρία Μπούχερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήλθατε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημαντική αυτή εργασία που κάνατε. Ελπίζω να συνεχίσετε. Γιατί η κοινωνία μπορεί να ωφεληθεί πολύ από το σημαντικό σας αγώνα κατά κάθε μορφή ρατσισμού κατά του αντισημιτισμού και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αυτό το project, αυτό το έργο να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες μορφές ε, ρατσισμού, για την καταπολέμηση, για παράδειγμα, του, των συναισθημάτων κατά των μουσουλμάνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να take ορίσουμε Begrüße ich herzlich την Ιντα Ερόλα και, την... και τον Βιλ Γιάρα που θα μας παρουσιάσουν το έργο Your European Citizenship, η ευρωπαϊκή σας ηθαγένεια, του Ευρωπαϊκού α, Κοινοβουλίου της Νεολαίας της Φιλανδίας. Δεύτερο βραβείο. So Εμείς εκπροσωπούμε ε, το, ε, την Ευρωπαϊκή Βουλή των Νέων ε, την Φιλανδία, της Φιλανδίας στα πλαίσια του, ε, της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Πρόκειται για μια μη πολιτική οργάνωση νέων Δεν υπάρχει τέτοιο κοινοβούλιο μονάχα στην Ευρώπη ε, και μονάχα στην Φιλανδία ε, και στην Αρμενία και στη Γεωργία ε, και σε άλλες χώρες και στη Σουηδία και την Νορβηγία υπάρχουν τέτοιου είδους κοινοβούλια. Ε, ε, στη διάρκεια των συζητήσεών μας ε, συζητούμε για πολιτικά ζητήματα, αλλά δεν έχουμε καμία υποστήριξη από πολιτικούς σχηματισμούς. Όλα οργανώνονται από νέους και για τους νέους και συνήθως ε, ε, όλοι όσοι ασχολούνται είναι ε, νέοι μέχρι 25 ετών. Εμείς λειτουργούμε σε όλη την Φιλανδία προσπαθώντας να οργανώσουμε εκδηλώσεις όχι μόνο στην πρωτεύουσα αλλά και σε άλλες πόλεις. Ε, εμείς έχουμε ένα project το οποίο περιέχει, περιλαμβάνει αρκετά ε, κεντρικά σημεία. Ε, πρώτα απ' όλα αυτό που ονομάζουμε school tours, δηλαδή η επαφή μας με τα σχολεία. Στα πλαίσια αυτά λέμε, βλέπουμε πώς μπορούμε να διαφημίσουμε κατά κάποιο τρόπο τη δράση μας στους νέους. Ε, ε, θέλουμε να οργανώσουμε ακόμα περισσότερα, περισσότερες εκδηλώσεις ε, στα σχολεία. χρησιμοποιούμε βέβαια πολύ και τα κοινωνικά δίκτυα και πλέον στις παρουσιάσεις που κάνουμε στα σχολεία, οι παρουσιάσεις αυτές έχουν γίνει ευρύτατες πλέον και παρουσιάζουμε όχι μονάχα τις δραστηριότητές μας, δεν διαφημιζόμαστε εμείς μόνο, αλλά προσπαθούμε να διευρύνουμε τη γενική γνώση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και την ε, Ευρώπη ε, και μέσω των παρουσιάσεών μας να παρουσιάσουμε και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ζωές μας και στις ζωές των πολιτών, αλλά και την σημασία της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Όπως είπαμε και προηγουμένως, εμείς κάνουμε εκδηλώσεις από νέους ε, για ε, νέους. Κάνουμε ε, τις παρουσιάσεις στα σχολεία σε όλη τη χώρα. Δεν έχουμε βέβαια πόρους έτσι ώστε να πάμε και σε σχολεία, σε πολύ μικρά χωριά, γιατί συνήθως οι εθελοντές μας προέρχονται από τις μεγαλύτερες πόλεις. τι κάνουμε στις ε, συνεδριάσεις μας. Ε, ε, οι συνεδριάσεις, στις συνεδριάσεις αυτές και στην ολομέλειά μας κάνουμε διεθνείς συναντήσεις όπου συμμετέχουν νέοι από όλη την Ευρώπη η κύρια ιδέα ε, είναι να γίνεται προσωμείωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, δηλαδή, στην αρχή οικοδομούμε ομάδες, team building δραστηριότητες, έτσι ώστε να γνωριστούμε μεταξύ μας και μετά συνεδριάζουμε σε επιτροπές, όπως είναι η Επιτροπή ε, το, της, του Πολιτισμού. Μπορεί να έχουμε και εμείς, δηλαδή, συνεδρίαση της Επιτροπής του Πολιτισμού και στα πλαίσια των διαφόρων επιτροπών συζητούμε τρέχοντα θέματα. Ε, και στο τέλος ε, συζητούμε ε, επί ψηφισμάτων και υπάρχει μετά η ψηφοφορία, είτε υιοθετεί, είτε εγκρίνεται, είτε απορρίπτεται το ψήφισμα. Να σας πω ότι Έχουμε και ε, ανθρώπους που έχουν γνωρίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, επί σειρά ετών και που μπορούν να συμμετάσχουν και να μας δώσουν τα φώτα τους. Και με τον τρόπο αυτό ε, συζητούμε τα θέματα όπως τα συζητάτε και εσείς στη πλαίσια των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους νέους, ε, γιατί δεν μαθαίνουν πολλά για την Ευρώπη στο σχολείο τους, ε, ε, όμως σιγά σιγά μαθαίνουν μέσα από τις δικές μας συνεδριάσεις και ενδιαφέρονται για την Ευρώπη. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε επίσης ανθρώπους να μάθουν αγγλικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Δεν μας ενδιαφέρει να μιλούν εξαιρετικά ή τέλεια αγγλικά, η διαδικασία διαδικασία μας ενδιαφέρει του ότι μαθαίνουν κάτι και κάνουν κάτι οι νέοι για τον εαυτό τους και για να αναπτύξουν την δράση τους και τις γνώσεις τους. Μετά από τις ε, συνεδριάσεις ε, δημιουργούνται φιλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχουν πλέον οι νέοι επαφές ε, σε με άλλες ε, χώρες, μπορούν να ταξιδέψουν έτσι ώστε να διοργανωθούν σιγά σιγά συνεδριάσεις και στο εξωτερικό. Ε, και βεβαίως επειδή μας ενδιαφέρει η διαδικασία μάθησης ε, ευελπιστούμε ότι κάθε συνεδρία θα ε, δώσει κάτι στους ε, συμμετέχοντες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ενθαρρύνουμε τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες, ε, ε, δηλαδή να είναι πραγματικοί πολίτες, ενεργοί, να έχουν μια ενεργή ηθαγένεια και αυτό να αρχίζουν να το μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία, πράγμα πολύ σημαντικό. Θα σας δώσω και κάποια αριθμητικά στοιχεία. Το 2018, λοιπόν, είχαμε τέσσερις συνεδριάσεις στη Φιλανδία και περίπου 500 συμμετέχοντες στη Φιλανδία. Κάναμε 24 παρουσιάσεις σε σχολεία και φέτος, μάλιστα, θα κάνουμε 50 παρουσιάσεις. Βλέπετε ότι έχουμε αύξηση. Ε, το 2018 είχαμε επίσης 40 διαφορετικές εθνικότητες που εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις μας, πράγμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για μας, σας δίνουμε τα στοιχεία μας ε, και μπορείτε να μας πείτε ενδεχομένως και τι κάνει το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ε, κάθε δική σας ε, χώρα, έτσι ώστε να εμπλουτιστούν και οι δικές μας γνώσεις. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας, λέει ο Πρόεδρος. ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμείς όλοι ως μέλη του Κοινοβουλίου γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να ε, γίνει γνωστή προς τα έξω η εργασία που κάνουμε στο Κοινοβούλιο. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν ε, συνειδητοποίησα ότι δεν είναι καθόλου γνωστή ε, ε, η εργασία μας. Το έργο μας είτε δεν είναι καθόλου γνωστό, είτε πολλοί κόσμος έχει πολύ ασφαλμένη αντίληψη για το έργο του Κοινοβουλίου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ακούγονται στο σχολείο οι εργασίες, στα σχολεία γενικά οι εργασίες του Κοινοβουλίου, γιατί διαφορετικά παραμένει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένας μέγας άγνωστος. Είναι πολύ σημαντικό σημαντική λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σας. Ωραία, συνάδελφοι, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε ερωτήσεις. Νίκολας. Ο Νίκλας. Έχω συμμετάσχει σε μία από τις ε, περιηγήσεις που κάνετε στα σχολεία, στη Γερμανία συγκεκριμένα. Το οποίο σημαίνει ότι είναι μια ιδέα που απλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Πολλοί άνθρωποι βέβαια δεν γνωρίζουν στην, ε, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στην ε, Ευρώπη και πώς λειτουργούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Έχουμε ένα πρόβλημα εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Οπότε η δουλειά που κάνετε εσείς είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί καλύπτεται ένα κενό που υπάρχει στο εκπαιδευτικό σύστημα στα κράτη-μέλη. Ένα κενό σε ό,τι την ύλη του προγράμματος. Ήθελα να σα ρωτήσω από πού χρηματοδοτήσετε και πώ μπορούμε να αυξήσουμε τη χρηματοδότησή σα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι το κάθε σχολείο στην Ευρώπη θα, έχει, θα συμμετάσχει σε αυτές τις σχολικές περιηγήσεις. Η χρηματοδότηση έρχεται από διάφορε πηγέ. Στη Φιλανδία, για παράδειγμα, το μεγαλύτερο τμήμα τη χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Παιδεία και πολιτισμού. Ε, έχουμε συνεργαστεί και με το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και ορισμένα μας, εκδηλώσει μας εκδηλώσεις χρηματοδοτούνται από το Erasmus+. Επίσης, υπάρχει το σχέδιο Understanding Europe, κατανοώντας την Ευρώπη. Δεν είναι το ακριβώς το ίδιο με εμάς. Ε, χρηματοδοτείται από την, το Ίδρυμα Schwarzkopf, και καλύπτει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα την Αυστρία και τις κάτω χώρες. Είναι ένα παρόμοιο σχέδιο με το δικό μας, παρόμοιο πρόγραμμα με το δικό μας. Εμείς ε, κάνουμε παρουσιάσεις μια ώρα στα σχολεία. Και ό,τι αφορά την χρηματοδότηση, σα είπα διάφορε πηγέ. Κυρίω το Erasmus Plus όμω και τα Υπουργεία είναι οι περισσότεροι, οι μεγαλύτερε πηγέ χρηματοδότηση. Ο κύριος Αντέμοφ. Συγχαρητήρια σε αυτούς τους νέους εδώ, που είναι πολύ χρήσιμο αυτό που κάνουν. Έχω κι εγώ συμμετάσχει σε τέτοιες πρωτοβουλίες ως δάσκαλος. Και στη χώρα μου την Βουλγαρία συχνά πηγαίνω από το ένα σχολείο στο άλλο και συναντώ τους μαθητές και τους μιλώ. Νομίζω ότι αυτές οι δραστηριότητες εντάσσονται στο Discover European Union, να καλύψει την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό να φτάσουμε στους πιο μεγάλους από τους μαθητές, πιο ηλικιωμένους από τους μαθητές, διότι είναι αυτοί οι οποίοι πιο γρήγορα θα φτάσουν να παίρνουν αποφάσεις. Χρειάζεται μεγαλύτερη πρόσβαση λοιπόν στην εκπαίδευση, περισσότερη δουλειά στην εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ και καλή σας επιτυχία. Δεύτερο βραβείο λοιπόν σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά σας και περιμένουμε κι άλλα νέα από εσάς. Thank you.

Αλίτσε Πλάτα και Φαμπιάνο Κατάνα από την Ιταλία. Σας καλωσορίζουμε. Γυροφώνικα. Αυτό είναι το πρόγραμμα που θα μας παρουσιάσετε, το οποίο και βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο. Έχετε το λόγο, κυρία Πλάτα, κυρία Κατάνια. Ε, Χαίρετε. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε για την δυνατότητα που μας δώσατε, το χρόνο που μας δώσατε, το βραβείο που μας απονείματε και το χρόνο κυρίως που μας δίνετε για να, να μιλήσουμε για το θέμα μας. Ε, εδώ και πολλά χρόνια ε, έχουν ξεκινήσει οι πανεπιστημιακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί κάποια κοινά ε, προγράμματα έτσι ώστε να ενεργοποιήσουν την ευρωπαϊκή νεολαία. Ακούσαμε και τα projects των συναδέλφων εδώ, των ε, άλλων βραβείων ε, ε, Καρλομάγνου και πραγματικά είδαμε πόσο σημαντικά είναι τα projects αυτά, αλλά και πόσες είναι οι πολλές δυσκολίες. Κύρια δυσκολία είναι το πώς μπορεί να φτάσει κανείς και να αγγίξει τους νέους της Ευρώπης. Εμείς ως ε, εκπρόσωποι ραδιοφωνικών ε, σταθμών των πανεπιστημίων αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το πάθος που έχουμε για τα μέσα ενημέρωσης έτσι ώστε να περάσουμε μηνύματα ε, πολιτισμού και ενεργοποίησης και δραστηριοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δημιουργήσαμε λοιπόν την Eurofónica. Πρόκειται για ένα project που αποτελεί για μας παράδειγμα των ραδιοφωνικών των σταθμών, των πανεπιστημιακών και των ε, όσων μπορούν να κάνουν οι νέοι. Τα college radios είναι ε, ιδιαίτερα μέσα ενημέρωσης γιατί ξέρουμε ότι το ραδιόφωνο είναι ένα από τα μέσα τα οποία ε, έχουν διαρκές, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από όλα τα υπόλοιπα μέσα αλλά λόγω των νέων τεχνολογιών, λόγω της τηλεόρασης, ε, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ, ε, οι πιο νέοι που ξεκινούν αυτήν την διαδικασία και που ζουν σε αυτήν την πραγματικότητα ε, βρίσκουν την ε, δυνατότητα ε, και να δώσουν μία διέξοδο στην ανάγκη επικοινωνίας τους, αλλά και να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Τα college radios είναι πολύ σημαντικά. Η οργάνωσή μας όμως λέγεται Ραντούνι. Είναι η οργάνωση δηλαδή των college radios στην Ιταλία και είναι ένα από τα συστατικά στοιχεία ε, της, ε, του project μας. Εμείς ε, οργανώσαμε, οργανωθήκαμε απέναντι στο βραβείο Καρλομάγνου ως ε, Ευρωφώνικα ε, της ε, Ιταλίας γιατί είχαμε την δυνατότητα εμείς να συνεδριάζουμε κάθε μήνα και αυτό δεν ίσχυσε για όλες τις άλλες εθνικές συνιστώσεις που δεν είχαν αυτήν την δυνατότητα. Εμείς έχουμε ραδιόφωνα λοιπόν που συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας, ραδιόφωνα τα οποία δημιουργούνται άμεσα στα πανεπιστήμια. Ε, και ε, στην Ιταλία όπως και σε πολλές άλλες χώρες ε, πρόκειται για καθαρά εθελοντικές οργανώσεις. Εμείς σε όλη μας την οργάνωση έχουμε μονάχα τους εθελοντές είτε στα College Radios είτε στην ευρωφωνιακά. Έχουμε 31 College radios στην Ιταλία και 300 μέλη ε, και ξέρουμε ότι και στις άλλες χώρες της Ευρώπης ε, είναι εξίσου ε, υψηλός ο αριθμός και πολλές φορές υψηλότερος ο αριθμός των συμμετεχόντων. Θα δώσω στον συνάδελφό μου τον λόγο για να μιλήσει για την Ευρωφώνικα. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε και η Αλίτσο, η Ευρωφώνικα είναι ένα project το οποίο δημιουργήθηκε, προέκυψε από την συνεργασία College Radios σε, από όλες τις χώρες χώρες. Ε, η Ραντούνη είναι μονάχα μία ε, από τις οργανώσεις ε, που συμμετέχουν. Έχουμε επίσης το Radio Campus France, το Άρου από τη Γαλλία, το Άρου από την Ισπανία, δύο από την Πορτογαλία ναι, και έχουμε επίσης ε, και συνεργασία με τα δίκτυα των Γερμανών και των Ελλήνων που δημιούργησαν τον αρχικό πυρήνα που οδήγησε μετά στην ε, Ευρωφώνικα. Η Ευρωφώνικα κατά την άποψή μας αντικατοπτρίζει την ε, σημασία της κατάρτισης, της πληροφόρησης, η ιδέα δηλαδή της εμπειρίας, της κατάρτισης και της δημιουργίας καθαρά ραδιοφωνικού περιεχομένου περιεχομένου, αλλά ε, και ε, που θα έχει στόχο την εξέβρεση νέων μοντέλων επικοινωνίας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το 2015 την Eurofónica, ε, η οποία μάλιστα δημιουργήθηκε μετά από μία πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς ξεκινούμε πλέον την πέμπτη περίοδο της Eurofónica ε, στην τελευταία περίοδο ε, έγινε μια μεγάλη αλλαγή. Από το 2015, όπως σας έλεγα και προηγουμένως και πάντα ε, λόγω της αρχικής μας τοποθέτησης απέναντι στον πειραματισμό που είναι το κυριαρχό μας όπλο, εμείς ξεκινήσαμε από το Vox Box περάσαμε ε, σε μια αλλαγή εποχή. Το Vox Box ήταν απευθεία σύνδεση με το Κοινοβούλιο, ε, ε, ενώ τώρα έχουμε 7 podcast την κάθε εβδομάδα. Και μια φορά τη βδομάδα κάνουμε και μια ανακεφαλαίωση της πολιτικής εβδομάδος που διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Χρησιμοποιούμε βεβαίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλες τις πλατφόρμες ε, που χρησιμοποιούν podcasting, firing ε, ε, και τα λοιπά που χρησιμοποιούν και οι νέοι. Από τη στιγμή της δημιουργίας της ευρωφώνικα. στόχος ήταν η πληροφόρηση για την Ευρώπη, για την διαδικασία πολιτικών αποφάσεων στην Ευρώπη, χωρίς όμως κάποια, κάποιο συσχετισμό με τα πολιτικά κόμματα στόχο ε, είχαμε πάντα τους νέους, όχι μόνο τους νέους ε, που βρίσκονται στα πανεπιστήμια, αλλά τους νέους γενικότερα από 30 και κάτω. Ε, νέους που θέλουν να ακούν ε, ραδιοφωνικό περιεχόμενο. Βεβαίως εμείς ε, προωθούμε τα περιεχόμενά μας κυρίως μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάνουμε λοιπόν αυτά τα podcasts και, καταλάβαμε ότι οι πλατφόρμες podcasting ήταν το καλύτερο μέσο ε, θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε και τα πανεπιστημιακά ραδιόφωνα ε, και γι' αυτό δημιουργήσαμε τα college radios σε όλη την Ευρώπη. Μετά περάσαμε ε, και στο βίντεο μέσα από τη χρήση της πλατφόρμας sitcom και άλλων που είναι πλατφόρμες μέσω Facebook. η Ευρωφώνικα πιστεύουμε ότι, ε, θα, ότι είναι ένα καλό παράδειγμα που ελπίζω να ακολουθηθεί και από άλλα, ένα καλό παράδειγμα έλεγα ε, πανεπιστημιακής συνεργασίας εμείς, συνεργασία με τους Γάλλους, με τους Ισπανούς ε, και άλλους φυσικά, ο καθένα στη γλώσσα του προστατεύοντας ε, και την διαφορετικότητα λοιπόν, είχαμε συνεργασία, συνεδριάζαμε, συναντιόμαστε κάθε μήνα στο Στρασβούργο και ε, δημιουργήσαμε λοιπόν αυτήν την ε, πλατφόρμα συνεργασίας από την οποία ε, θα μπορούσαν να απορρεύσουν η οροφόνικα Ιταλίας, η οροφόνικα Γαλλίας κλπ. Κοιτάξτε, ε, ο καθένας ακολουθεί το δικό του ε, πανεπιστημιακό ε, πεδίο. Μπορεί να γίνει γιατρός, μπορεί να ασχοληθεί με μέσα ενημέρωσης, αλλά όλοι μπορούν να ασχοληθούν ε, με το ραδιόφωνο. Έτσι συνεργάζονται και συναντιούνται διαφορετικοί τομείς, διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικοί πολιτισμοί αυτοί που μιλούν περισσότερες γλώσσες ε, βοηθούν έτσι ώστε η μετάφραση να γίνεται σε όσο γίνεται περισσότερες γλώσσες και έτσι ώστε ε, το κοινό μας να δέχεται το μήνυμα στην μητρική του γλώσσα. Ε, καταλαβαίνετε όμως ότι βλέπουμε το θέμα και από το, την οπτική γωνία των διαφορετικών ενδιαφερόντων. Έχουμε ανθρώπους γιατρούς, μεταφραστές, ε, αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με τη βιολογία, με την ευρωπαϊκή πολιτική ή τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Μιλάμε λοιπόν για συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικούς ε, τομείς, πράγμα που σημαίνει ότι ε, συζητούμε τα θέματα, γιατί πριν τα εκφράσουμε προς τα έξω, βεβαίως τα συζητούμε συζητούμε μεταξύ μας. Άρα διεθνή συνεργασία ε, ε, όσον αφορά ορισμένα θέματα και προσέγγιση διαφορετικών κοινών. Όπως έλεγε και ο συνάδελφος προηγουμένως, εμείς απευθυνόμαστε ε, σε φοιτητέ, σε ανθρώπους που είναι κάτω των 30 ή που είναι ακόμα, ε, όμως διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να ακουμπήσουμε και ε, κοινά τα οποία είναι ακόμα, παιδιά τα οποία είναι ακόμα στο Λύκειο ή και ευρύτερο κοινό όπως είναι οι μητέρες μας, οι γιαγιάδες μας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί εμείς φιλοξενούμεθα από εσά στο Στρασβούργο, χρησιμοποιούμε ε, τα ραδιοφωνικά στούντιο ε, της, ε, του, του Στρασβούργου και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς καταλαβαίνουμε αυτό που συμβαίνει έτσι ώστε να το μεταφέρουμε στους άλλους. Τα college radios είναι πολύ σημαντικά με την έννοια ότι παράγουν είναι πολύ σημαντικό το περιεχόμενο που παράγουν. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μετάδοση σε 24ωρη βάση και τα περιεχόμενα μπορεί να διαφέρουν πάρα πολύ. Αυτό που θέλουμε και αυτό που λέμε πάντα είναι ότι ήρθαμε σε επαφή με την Ευρώπη αλλά το σλόγγαν μας είναι ενωμένοι στη διαφορετικότητα, δηλαδή δεν θέλουμε να γίνουμε όλοι οι ίδιοι. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, είναι πολλά ε, τα προγράμματα τα οποία μπορούν να φτάσουν ε, μέχρι τους νέους, ε, να γνωστοποιηθούν στους νέους μέσα από το ραδιόφωνο με μικρό κόστος. Και να προσθέσω κάτι αν μου δίνετε τη δυνατότητα, κάτι ιδιαίτερο και να πω ότι η πρώτη συνέντευξη που κάναμε ήταν στον Ντάβιντε Σασόλη πριν γίνει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να παίξετε το βίντεο σας παρακαλώ.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 Thank you very much for coming. And... Ευχαριστώ. Σας συγχαίρω και πάλι για το πρώτο βραβείο το οποίο το αξίζετε. Σας ευχαριστώ για τη δεσμευσή σας και ελπίζουμε να συνεχίσετε τις εργασίες σας. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Κυρία Σόιτροβα. I, I know that we are very... Ξέρω δεν έχουμε πολύ χρόνο, συγχαρητήρια όμως για αυτό το βραβείο. Στην παρουσίασή σας απάντησατε σχεδόν όλες μου τις ερωτήσεις. Ε, αλλά να σα ρωτήσω το εξή Και εργάζεστε και σπουδάζετε ταυτόχρονα. Αυτή είναι η μόνιμη ερώτηση. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. E Είμαστε οι περισσότεροι από εμά ε, ε, φοιτητές, αλλά ε, έχουμε και τους λεγόμενους αλούμνοι, ε, τους αποφύτους που παραμένουν στην διαδικασία έτσι ώστε να περάσουν την τεχνογνωσία και στους επόμενους φοιτητές. Ξέρετε ότι όμως και πολλοί από εμά παραμένουν στο Πανεπιστήμιο. Εγώ εργάζομαι πλέον στο Πανεπιστήμιο. Ξεκίνησα λοιπόν το Πανεπιστημιακό Ραδιόφωνο ε, και τώρα συνεχίζω μια και εργάζομαι πλέον στο Πανεπιστήμιο. Eh. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί αγαπητή Αλίτσε, ε, λέει ο κύριο Μερίλιο, αγαπητέ Φαμπιάνο, είναι εξαιρετική η δουλειά επικοινωνίας και πληροφορίας ελεύθερης ε, που κάνετε. Ε, πραγματικά δημιουργείται μία δικτύωση, όχι μόνο σε επίπεδο Ιταλικών Πανεπιστημίων, μία δικτύωση όμως η οποία έχει σαν κύρια στοιχεία την αυτονομία. Πρέπει να πω ότι ο Αντώνιο Μεγαλίτσι, ένα νέο δικό μα άνθρωπο άνθρωπος ε, ο οποίος πραγματικά έκανε αυτή τη δουλειά, ε, δολοφονήθηκε στο Στρασβούργο ε, την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω ότι πρέπει να μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο και περισσότερο για σας. Εμείς είχαμε παρουσιάσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο δυστυχώς και περιέργως δεν έλαβε την απαραίτητη πρόθεση δεν και έγκριση. Γι' αυτό θα πρέπει να μας πείτε πώς είναι δυνατόν να βοηθήσουμε έτσι ώστε διαρθρωτικά να βοηθήσουμε <coughs> την Ευρωφώνικα και επίσης να μας πείτε και πώς από εθνικό ιταλικό project έγινε ένα project ε, ευρωπαϊκό ή πώς μπορεί να γίνει ακόμα πιο ευρωπαϊκό. Ναι, και εγώ θα ήθελα ε, να πω ότι ο, πραγματικά ο Αντώνιο Μεγκαλίτσι ήταν στο Στρασβούργο στα πλαίσια της δικιάς μας ε, διαδικασίας. Ήταν στην ε, ε, ε Ευρωφώνικα, αλλά ε, πραγματικά θα ήθελα να ε, υπενθυμίσω και να θυμίσουμε και να θυμηθούμε και όλους τους άλλους ε, που υπήρξαν θύματα. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν σχέση και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντως ήταν μια στιγμή η οποία πραγματικά χαράκτηκε στη μνήμη και στη συνείδηση των Ευρωπαίων. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα δίκτυο των πανεπιστημιακών ραδιοφώνων στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ε, και ε, Τώρα, για το πώς μπορούμε να ε, δουλέψουμε περισσότερο. Το πρώτο θα ήταν να κινητροδοτηθούν τα εθνικά γραφεία εκπροσώπησης του Κοινοβουλίου και έτσι ώστε να βοηθηθούν οι νέοι, κυρίως όσον αφορά τα ταξίδια ε, που κοστίζουν ε, πολύ. Εμείς είχαμε μια καλή επαφή ε, με, την, με το γραφείο του Κοινοβουλίου στην Ιταλία. Στην ουσία όμως εμείς οι ίδιοι οι νέοι, οι speaker του ραδιοφώνου που βάζουν τα χρήματα για τα ταξίδια ε, και ε, επίσης σε εθνικό επίπεδο έχουμε και κάποια συνεισφορά ε, η οικονομική η οποία μας βοηθάει. Αλλά αν θέλετε να μας βοηθήσετε ε, ακριβώς μέσα από τα προγράμματα της Δημιουργικής Ευρώπης θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε. Εμείς, ε, όπως, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ε, είχαμε υποβάλει ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο δεν έγινε δεκτό. Τώρα, υπάρχει ένα πρόβλημα με τις γλώσσες. Ε, και με την έννοια του έργου ε, το περιεχόμενο της ραδιοφωνικής εκπομπής δεν θεωρείται έργο ε, καλλιτεχνικό. Εμείς ζητούμε να ενταχθούμε στη Δημιουργική Ευρώπη γιατί βάσει του project των των ε, ραδιοφώνων των πανεπιστημιακών εμείς μιλάμε για πάρα πολλά θέματα, για κινηματογράφο, για ε, διατροφή, για ιατρική, ε, ιατρικά θέματα κλπ. Εάν αυτό δεν είναι ευρωπαϊκή δημιουργία, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nur noch... Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να δούμε τα διάφορα. Για τη δημόσια κρέαση, η κυρία Μπεντζομέρ έχει ένα σχόλιο να κάνει. Παρακαλώ. Gracias, presidente. Sí, muy brevemente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καταγγείλω εδώ σε αυτή την Επιτροπή την ε, πολύ σοβαρή κατάσταση η οποία επικρατεί στην Καταλωνία στα πανεπιστήμια. Εκεί οι Πριτάνης και τα Πριτανικά Συμβούλια κρατικών πανεπιστημίων έχουν αποφασίσει να ξεχάσουν το καθήκον τους τα πανεπιστήμια να είναι χώροι ελευθερίας και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα όργανα αυτά για λόγους πολιτικούς και ιδεολογικούς, στηρίζοντας ομάδες φοιτητών που διοργανώνουν διαμαρτύριες που έχουν ως αποτέλεσμα χιλιάδες ε, ε, Ισπανών φοιτητών στην Καταλωνία να μην μπορούν πλέον να ασκήσουν το δικαίωμά τους ε, να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, να συμβιώσουν ελεύθερα και να αξιολογούνται. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχει το φόρουμ των Ισπανών πανεπιστημιακών καθηγητών για την συμβίωση, οι οποίοι καταγγέλουν την κατάσταση αυτή και τη στάση των Βρετάνων και των Βρετανικών Συμβουλίων. Ευχαριστώ. Äh, Είναι σημαντικό το θέμα αυτό, το οποίο δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να το εξετάσουμε σήμερα. Θα πρότεινα να μπει στην ημερησία διάταξη των επόμενων συνεδριάσεων προκειμένου να το συζητήσουμε. Και τώρα να περάσουμε στο, στους τριμερείς διαλόγους, το ε, τελευταίο σημείο στην ημερησία διατάξη της σημερινής συνεδρίαση. Και αυτό θα γίνει και κλεισμένο το θηρόν το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να καλέσω όλους τους παραβρισκόμενους που δεν είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να βγουν από την αίθουσα. Ευχαριστώ.